Buongiorno, Καθίστε, αρχίζουμε αμέσως. Ας δώσουμε μερικά δευτερόλεπτα στους συναδέλφους για να καθίσουν. Έλεγα ότι αρχίζουμε αμέσως και ρωτώ εάν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη όπως έχει. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται κατά συνέπεια η σε διάταξη. Πρέπει να εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά της 17ης-18ης Σεπτεμβρίου 2012, 24 Σεπτεμβρίου 2012, 15 Οκτωβρίου 2012. Και εδώ αν δεν έχετε αντιρρήσεις θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Πριν ξεκινήσουμε την ακρόαση σας θυμίζω ότι η συνεδρίαση αναμεταδίδεται απευθείας από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσουν και κλεισμένων των θυρών οι συντονιστές της Επιτροπής. Ξεκινάμε τις ακροάσεις μας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις μέρες ε, αποστολή στην Ιταλία και έχουμε διάφορα κεφάλαια. Πρώτον είναι προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Θα ακούσουμε το Τόμ Νίλαν που είναι ε, από τη γραμματεία της FATF. Μετά ο Ούγκο Μπάση, ο διευθυντής στην DG, στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς θα μας παρουσιάσει ένα αντίστοιχο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της FATF. Δέκα λεπτά για κάθε παρουσίαση, δύο λεπτά ο κάθε βουλευτής, πρώτα οι συντονιστές και μετά οι εισηγητές. Μετά θα απαντήσουν οι εισηγητές και άπαξ και έχουμε χρόνο θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πληροφορήσω ότι ο συνάδελφος Κροτσέτα από το, την προηγούμενη εβδομάδα είναι πλέον κυβερνήτης της Σικελίας. Τον παρακάλεσα να έρθει σήμερα, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να έρθει, αλλά σας παρακαλώ να προχωρήσουμε στην εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο δόκτωρ Τόμ Νίλαν από τη γραμματεία της FATF. Ο δόκτωρας, δόκτωρα Νίλαν, έχετε 10 λεπτά. Και μετά ο δόκτωρ Μπάση θα μιλήσει. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα γνωρίζετε ότι η FATF είναι Διεθνής ε, Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και θέτει τα πρότυπα. Έχουμε 40 συστάσεις αλλά μόλις 10 λεπτά. Ε, κατά ανάγκη λοιπόν θα είμαι πάρα πολύ επιλεκτικός. Το πρώτο που θέλω να πω είναι λίγο το ιστορικό υπόβαθρο. Γιατί έχουμε αυτά τα πρότυπα της FATF. Ε, η νομιμοποίηση εσόδων από εκκληματικές δραστηριότητες είναι ε, σημαντικό ποσοστό του παγκοσμίου ΑΕΠ και Βεβαίως ένα πολύ μικρό ανακαλύπτεται ε, ε, με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ ε, για τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα. Βλέπουμε το πρόβλημα είναι μεγάλο. Τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά μέτρα είναι σχετικά αποδοτικά μπορούμε να βρούμε ποια είναι η εγκληματική δραστηριότητα ε, που αποφέρει ε, έσοδα, είναι 70% Έχουμε την επιβολή του νόμου αλλά και άλλες μορφές, ειδική ε, πληροφόρηση για τα οικονομικά. Η δίμευση, η κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος είναι πολύ ε, μεγάλος αποτρεπτικός παράγων. Επίσης ε, και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης βοηθάει για να είναι το περιβάλλον εχθρικό προς τους χρήστες αυτούς για να προστατεύεται τελικά το χρηματοοικονομικό σύστημα από παράνομα έσοδα και να προστατεύεται και η ακαιρεότητά του. Η Ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης στήθηκε το 1989 για να καταπολεμήσει το ξέπλυμα ε, του χρήματος που συνδέεται κυρίως με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Χρειάστηκε τότε να συντονιστεί αυτή η δράση. Η εντολή μας έχει διευρυνθεί και από το 2001 αντιμετωπίζει και την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και από φέτος και ε, τη χρηματοδότηση της διάδοσης ε, όπλων μαζικής ε, καταστροφής. Εργαζόμαστε ως ειδική ομάδα Task Force. Δεν έχουμε εντολή με βάση τον νόμο. Είναι θελούσια η εφαρμογή των συστάσεών μας. Ωστόσο, είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό που ονομάζεται Διεθνές Ήπιο Δίκαιο. Γιατί είμαστε τόσο αποτελεσματικοί. Έχουμε πρότυπα, όπως σας είπα, και ένα μηχανισμό αξιολόγησης, σύγκρισης ομοτήμων μεταξύ ε, κρατών ε, για να δούμε αν συμμορφώνονται και πώς ε, εξασφαλίζεται η ακαιρεότητα του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος. Βλέπουμε, ας πούμε, ποιες χώρες δεν έχουν τα σωστά συστήματα και καταρτίζουμε και ε, μαύρους καταλόγους, μαύρες λίστες για τις χώρες που προσφέρονται για ξέπλυμα. Οι 40 συστάσεις μας το τελευταίο διάστημα αναθεωρούνται για να βελτιωθεί ε, το σύστημα καταπολέμησης νομιμοποίησης όδων από εγκληματικέ δραστηριότητες. Βλέπουμε ποιες είναι οι αδυναμίες και ε, θέλουμε να ενημερώσουμε το σύστημα για να δούμε και ποιες είναι οι σύγχρονες πρακτικές στο χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτό γίνεται ανάμεσα στους διάφορους γύρους ε, ελέγχου μεταξύ των διαφόρων κρατών. Ε, με την Ισπανία θα αρχίσουμε το επόμενο διάστημα, τον επόμενο γύρο, τον Ιανουάριο του 2014. Εξετάζουμε λοιπόν τα εθνικά συστήματα για να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι και όχι τόσο πολύ ε, αν ανταποκρίνονται τεχνικά και θεσμικά και νομικά οι μηχανισμοί του κράτους. Βλέπετε εδώ την οθόνη με τα μέλη μας, 34 κράτη-μέλη δύο περιφερειακές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ε, ξεχωριστό μέλος. Έχουμε και 14 ε, κράτη-μέλη της Ένωσης που είναι μέλη μας. Ε, εκτός αυτού έχουμε και 8 περιφερειακούς οργανισμούς που μας υποστηρίζουν, όπου συμμετέχουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και λίγα είναι τα σημεία του κόσμου που δεν καλύπτουμε και προσεχώς θα τα καλύψουμε και αυτά. Ποια είναι τα βασικά θέματα που καλύπτουν τα πρότυπα και οι προδιαγραφές μας. Ό,τι έχει να κάνει με ένα αποτελεσματικό εθνικό σύστημα για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν θα μπω ε, σε λεπτομέρειες, αλλά αυτά τα θέματα και οι τομείς υποστηρίζουν ένα τον άλλον στο ποινικό δίκαιο ας πούμε και το ποινικό σύστημα των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζονται και προληπτικά μέτρα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε κάποια άλλα επαγγέλματα ή επιχειρήσεις όπως είναι τα καζίνο ας πούμε. Θα πρέπει επίσης να ελέγχονται αυτές οι υποχρεώσεις ως προς την τήρησή τους, να υπάρχουν αρχές για τη ε, διαχείριση και τη συλλογή ε, πληροφοριών για ύποπτες δραστηριότητες οικονομικής φύσεως, ειδικά μέτρα ε, για την ε, διαχείριση κάποιων στοιχείων ενεργητικού ε, εταιριών όπως είναι τα αυτοκίνητα. Και τώρα στην πολιτική και το συντονισμό είναι πάγια η απέτηση να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών. Ε, είναι πολλοί οι κρατικοί φορείς που πρέπει να συνεργάζονται στο θέμα του ξεπλήματος χρήματος. Βλέπετε το κείμενο ε, με ε, κόκκινο για το τι θα γίνει φέτος για την αναθεώρηση των προδιαγραφών. Ε, βάζουμε, θέτουμε την έμφαση περισσότερο στην προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, το ρίσκο. Για πρώτη φορά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εντοπίζουν ποιους κινδύνους διατρέχουν ειδικά οι χώρες και να τις αξιολογούν και να λαμβάνουν το υπόψη όταν ε, θέτουν, ε, θεσπίζουν κανόνες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή όταν επανεξετάζουν το θέμα της διάθεσης των πόρων σε διάφορους μηχανισμούς και θεσμούς του κράτους. Θα πρέπει οι να κατανοούν τον κίνδυνο. Αυτό Τώρα μόλις αρχίζουν να το καταλαβαίνουν ορισμένε χώρες. Έτσι όμως γίνεται το σύστημα ακριβώς πιο αποτελεσματικό για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του χρήματος ε, και ελαφρύνεται ο πιστοτικός τομέα και κάποια επαγγέλματα χαμηλού ρίσκου αρκεί να, τον εντοπίσει κανείς τον κίνδυνο για να καταλάβει που πρέπει να δράσει. Ε, η νομιμοποίηση εισόδων λοιπόν από εγκληματικές δραστηριότητε και η δίμευση κατάσχεσή του είναι το βασικό μα έργο. Ε, θέλουμε να ποινικοποιείται αυτή η δραστηριότητα και να δημεύονται τα ε, περιουσιακά στοιχεία των ε, εγκληματιών και βεβαίω να εφαρμόζονται αυτά. Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή από φέτος. Τα φορολογικά εγκλήματα προστίθενται στον κατάλογο των ποινικοποιούμενων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πολλά κράτη ήδη το κάνουν. Λίγες είναι οι χώρες που χρησιμοποιούν κατάλογο ε, αξιόπινων πράξεων που ορίζουν ακριβώς τι νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητε. Έχουμε τα πρότυπά μας και τις προδιαγραφές μας, αλλά οι χώρες που στο παρελθόν δεν ακολουθούσαν αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να παρέχουν διεθνή συνεργασία προς άλλες χώρες που θέλουν να διερευνήσουν εγκληματικέ πράξεις που σχετίζονται με το φορολογικό έγκλημα και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Αυτό ε, έχει ενδεχομένως ε, σημασία, αλλά είναι αρκετά περιορισμένο το πεδίο. Ε, τώρα, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης ε, των όπλων μαζικής καταστροφής. Είναι ήδη μηχανισμοί με το ξέπλυμα χρήματος, αλλά έχουν και επιπλέον ειδικά της τρομοκρατίας. ζητούμε από τις χώρες να ποινικοποιήσουν βεβαίως τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με ειδικέ κυρώσει, όπω προβλέπεται από το Συμβούλιο Ασφαλεία των Εθνών, και ειδικά μέτρα και ασφαλιστικέ ε, δικλείδε για τα κέρδη. Ποια αλλαγή κάναμε φέτος. Ε, προσθέσαμε τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής με μια νέα σύσταση έτσι ώστε να ε, γίνεται πιο σωστή και πιο αυστηρή εφαρμογή των μέσων ε, και των κυρώσεων που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο ασφαλεία του ΟΗΕ, ιδιαίτερα για το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Είναι πολύ περιορισμένο το πεδίο εφαρμογή εδώ, δεν προσθέτει τίποτα στι απαιτήσει του ΟΗΕ, αλλά είναι σημαντικό ε, ακριβώς ε, το ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή αυτό το μέτρο. Τώρα έρχομαι στα προληπτικά μέτρα. Αυτά ζητούνται από κάποια επαγγέλματα και από τις τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το σημείο εισόδου των χρημάτων αυτών στο χρηματοοικονομικό σύστημα, να ε, προσδιορίζεται η ταυτότητα του προσώπου που προβαίνει σε αυτή τη δραστηριότητα και ποια είναι η οικονομική συναλλαγή. Υπάρχουν και άλλες απαιτήσει για τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εμβάσματα και ροές χρηματικές. Από φέτος το Φεβρουάριο έχουμε διευρύνει ε, τις απαιτήσει ε, για ε, προβεβλημένα πολιτικά πρόσωπα άλλων χωρών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων κτλ. Τώρα αφορά και κάποια άλλα πρόσωπα και πολιτικούς, όχι μόνο τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και αλλού στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν οι πιο αυστηροί κανόνες πλέον που αφορούν τα νομικά πρόσωπα και τα ε, αυτοκίνητα των εταιριών. Εδώ και καιρό το ζητούμε γιατί υπάρχει κατάχρηση ε, σε κάποιους ομίλους και σε κάποιες εταιρείες αλλά δεν ήταν ε, αρκετά ικανοποιητική εφαρμογή. Κάνουμε λοιπόν νέες συστάσεις πολύ πιο λεπτομερείς για το τι θα πρέπει να κάνουν οι χώρες για να καταπολεμήσουν την κατάχρηση τέτοιων φαινομένων. Πρώτο τελευταίο στοιχείο. Ποιε είναι εξουσίε των αρμοδίων αρχών. Ε, ανακριτικές εξουσίες, ε, ερευνητικέ εξουσίες, ε, επιτήρηση και άλλα τεινά που πρέπει να έχουν αρχές επιβολής του νόμου. Αυτά ήταν παλιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα φέτος. Στις αρχές όμως του 2012 εγκρίναμε νέες συστάσεις για να αρθούν ορισμένα πρακτικά εμπόδια που δεν ε, καθισούσαν δυνατή τη συνεργασία των κρατών ε, το τελευταίο διάστημα. Παραμένουν ήδη σε αρχές, αλλάζουν όμως τα πρακτικά εμπόδια και καταργούνται. Αυτή είναι η σύνοψη. Ήταν πάρα πολύ ε, μικρή και βραχή επισκόπηση για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές για μας και τα κράτη-μέλη μας, τώρα η εστίαση ποια θα είναι. Αυτές οι αλλαγές που έχουν είναι να μεταφερθούν με τρόπο αποτελεσματικό στο εθνικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δόκτωρα Νίλαν. Ο δόκτωρο Ούγκο Μπάσια έχει το λόγο, ο οποίος είναι διευθυντής της Digimart της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε κυρία Αλφάνο, θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Πρώτα απ' όλα, κατά τη διάρκεια της σύντομης παρέμβασής μου, θα ήθελα βασικά να κάνω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να σας πω αυτό το οποίο μπορώ τώρα να σας πω για την συνεσυζόμενη διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου για την, ε, στην Ευρώπη για την καταπολέμηση των ε, ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Σύντομα θα έχουμε μία νέα πρόταση, κυρίως για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις νέες αρχές έτσι όπως έχουν τροπολογηθεί από φέτος το ε, Φεβρουάριο. Πρόκειται για τις συστάσεις της FA της F και να σας πω επίσης ποια είναι η πολιτική που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις αλλαγές εκ μέρους της Επιτροπής ώστε να είμαστε σίγουροι το νέο σύστημα θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά στην ενιαία εσωτερική αγορά. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να τονίσω πόσο σημαντική είναι η εργασία που επιτολεί η Επιτροπή σας, που έχει μεγάλη σχέση με αυτά τα οποία κάνει η FATF και εμείς, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο. Θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να συνεργάζονται μαζί, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα θα πρέπει να κάνουν μια συμπληρωματική προσπάθεια, διότι, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Τόμα, μιλούμε για ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τα αποτελέσματα και επιπτώσεις των πρώτων προσπαθειών που καταβλήθηκαν και παγκοσμίω και σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο. Πρέπει να πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ενθαρρυντικά, αλλά βλέπετε ότι είναι τρομακτική αριθμή και μπορώ να προσθέσω και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλέστηκε και ο τα ποσά τα οποία ταυτοποιούνται, εντοπίζονται, είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση με το σύνολο του κεφαλαίων τα οποία παγκοσμίως ε, περνάνε από αυτή την παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να διαδρομητήσουμε συμπληρωματικέ προσπάθειες και είμαστε έτοιμοι εμεί να παίξουμε το ρόλο μα. Ο ρόλο τη FATF βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμμετέχουμε στι εργασίε και συνεργαζόμαστε και εν παραλίλω με την FATF και πιστεύουμε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να εξασφαλίσουμε το ότι θα έχουμε υψηλού επίπεδου προδιαγραφές οι οποίες στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας θα εφαρμοστούν εναρρονισμένο. Όπως σας είπα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι αρχές εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι αυτό το οποίο κάνουμε εργαζόμενοι για την ε, αναθεώρηση της οδηγίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και βεβαίως έχουμε το, την ειδική πρόκληση στην ενιαία εσωτερική αγορά. Δηλαδή, όπως σας είπα, ενεργούμε στην ενιαία εσωτερική αγορά όπου πρέπει να συνεχίσουν να συνεχούμε να εγγυόμεθα κάποιες ελευθερίες, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, ελεύθερη κυκλοφορία τόμων και υπηρεσιών. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να επιβάλλουμε ελέγχους δυνητικά ε, για να μειώσουμε αυτή την ελευθερία θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ την ελευθερία αυτή που παρέχεται από την ενιαία εσωτερική αγορά και την αποδοτικότητα των ελέγχων που επιβάλλουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολύ σημαντικούς στόχους όπως αυτόν για τον οποίο μιλούμε σήμερα. Γι' αυτό πρόκληση και εργασία μας δεν είναι εύκολη και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε ειδικέ προκλήσεις. Όταν πρόκειται βεβαίως στο κοινωτικό δίκαιο να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές. Προσπαθούμε παρόλα αυτά και αυτό το οποίο προσπαθούμε να ε, εφαρμόσουμε και να το εφαρμόσουμε στο νέο πλαίσιο και σύντομα θα έχουμε μπροστά μας μία πρόταση της Επιτροπής θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ελπίζουμε, προς έγκριση. Το κύριο στοιχείο αυτού του νέου καθεστώτος θα είναι η αλλαγή από μία ε, προσέγγιση όπου προτείνουμε μέτρα, σε μία προσέγγιση όπου τα μέτρα θα βασίζονται στον κίνδυνο, στο ρίσκο που υπάρχει. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε πιο εστιασμένη, πιο στοχευμένη προσέγγιση στους κινδύνους. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι η ευθύνη όλων των εμπλεκομένων και των φορέων που στους διάφορα επίπεδα ε, είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κανόνων, θα αυξηθεί και από την προσέγγιση την, ε, του tick box την ημιαυτόματη ε, θα είναι πιο στοχευμένη. Πιστεύουμε ότι θα πρόκειται με τον τρόπο αυτό για μια πολύ μεγάλη βελτίωση και θα μας επιτρέψει να εξοικονομήσουμε και πόρους από την άλλη. Δεν είναι μόνο τον, το μοναδικό στοιχείο το οποίο θέλουμε με στα πλαίσια των αλλαγών που θέλουμε να κάνουμε στο σύστημα που ισχύει. Σε κάποιους τομείς θα προχωρήσουμε περισσότερο και από τις αρχές της FATF θέλουμε να επεκτείνουμε το ε, των αρχών αυτών και των φορέων και των δραστηριοτήτων που θα καλύπτει ενδεχομένως η νέα νομοθεσία. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, θέλουμε να καλύψουμε και τα παιχνίδια, τα παίγνια και όχι μόνο τα καζίνα όπως αναφέρεται στις τάσεις της FATF. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το ειδικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε κάποιες έννοιες, να εισαγάγουμε το στοιχείο της διαφάνειας όσον αφορά τους ορισμούς, όσον αφορά τον πραγματικό δικαιούχο, θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, διαφάνεια. Τώρα, οι κυρώσει. Το σύστημα κυρώσεων θέλουμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό, διότι αν δεν εφαρμόζεται σωστά ο κανόνα και δεν υπάρχουν κυρώσει, είναι άχρηστο να εφαρμόσουμε ένα νέο καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε το ότι οι κυρώσει θα πρέπει να είναι αυτές που χρειαζόμαστε και γενικά προσπαθούμε να είμαστε γενικότερα και σε όλους τους τομείς πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί. Κυρίως εξασφαλίζονται ότι τα κράτη-μέλη όχι μόνο θα διαθέτουν την κατάλληλη νομοθεσία, αλλά ότι θα μπορέσουν να την εφαρμόσουν και με τον σωστό τρόπο. Βεβαίως, αν αυτό είναι κυρίως θέμα των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, προσπαθούμε εμείς να δώσουμε την ΕΣΜΑ και περισσότερες αρμοδιότητες, ώστε όχι μόνον οι ορισμοί, οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν το σχετικό δίκαιο να ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά διασφαλίζοντας ότι θα μπορέσουμε να ε, επέμβουμε και σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες από τις εθνικές αρχές. Τελικά, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τον αριθμό και την ποιότητα των μέσων, των εργαλείων που θα διαθέσουμε και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο φαινόμενο. Και όπως είπα, επεξεργαζόμαστε την πρόταση. Η μελέτη επιπτώσεων ολοκληρώνεται και θα παρουσιαστεί μαζί με την πρόταση. Προσπαθούμε να χτενίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και σύντομα θα ολοκληρωθεί Πολύ δύσκολο βεβαίως να αναφέρω τις ε, ημερομηνίες έγκρισης, αλλά σύμφωνα με το παρόν χρονοδιάγραμμα, η έγκριση της πρότασης πιστεύουμε ότι θα γίνει τους πρώτους μήνες του επομένου έτους. Και βεβαίως όταν υποβληθεί η πρόταση στα νομοθετικά όργανα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να συνεργαστούμε αποδοτικά όπως συνήθως και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε το πλαίσιο κανόνων αυτών να το έχουμε στη διάθεσή μας έτοιμο στο τέλος του 2013. Πρόκειται για κάτι το ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Και 20 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσω θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στην Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ξεκινάω τώρα τη συζήτηση. Δύο λεπτά ο κύριος Γιακολίνο που είναι εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω κι εγώ να κρατήσω το χρόνο μου. Όπως έπραξαν και οι δύο εισηγητές. Για το θέμα της ανακύκλωσης που συνδέεται με την διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα για το οποίο συζητήσαμε και στην Ιταλία τις προάλλες στην αντιπροσωπεία. Υπάρχει ένα θέμα χωρών που βρίσκονται σε μία μαύρη λίστα. Και υπάρχει ένα θέμα που δεν έφυξε ο κύριος ο εισηγητής ε, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών. Εμείς πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν την νομοθεσία όπως πρέπει. Τώρα για την ε, τελευταία τοποθέτηση έχουμε μια, εδώ μια προσέγγιση περισσότερο για τα ρίσκα και όχι για τις υποχρεώσεις. Μπορείτε να είστε ακριβέστερος κύριε Διευθυντά. Και μια άλλη ερώτηση για την αυτοανακύκλωση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά, σε άλλους όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα με έναν ενιαίο κανόνα, δεν θα ήταν χρήσιμο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο, οι Κύριο Σπαγιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο εμπειρογνώμονες για τις ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Μερικές παρατηρήσεις μόνο σε σχέση με τη σημερινή ακρόαση για την νομιμοποίηση έσοδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος των χρημάτων που διακινούνται. Υπάρχουν και στοιχεία από τα Ηνωμένα Έθνη. Το 2009 Ε, αυτό υπολογίζεται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το έδειξε και η οικονομική κρίση, ότι πρόκειται για ένα είδος εγκλήματος που ε, αφορά μεγάλες τράπεζες. Το έχει αναφέρει και ένας Ιταλός συγγραφέας, ένα πολύ γνωστό του ε, βιβλίο, Ρομπέρτο Σαντιάνο, και ε, μιλάει για 200 με 700 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε αυτά που μας λέτε, τονίσατε ότι θα πρέπει να καταλάβουν τα κράτη-μέλη την απειλή που συνιστά το ε, ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματος. Γιατί δεν το αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη. Εσείς έχετε κάποια δυνατότητα σύγκρισης. Το μετράτε αυτό, με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη τα εφαρμόζουν, τα μεταφέρουν στην νομοθεσία τους, αυτά που εσείς ε, τους συνιστάτε στη χώρα μου, τη Σλοβενία, γίνεται συζήτηση αυτό το καιρό σχετικά με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλλονται. Όταν αποκαλύπτονται αυτά, μπορεί να αυξηθεί και η συλλογή φόρων και βρίσκεται ε, σε Παρασκευή τώρα ένα νομοσχέδιο να αποκαλύπτεται το όνομα μεν ε, των ε, προσώπων αυτών, αλλά όχι το ποσό. Τι να το κάνουμε αυτό. τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αν κάποιο, α πούμε, έχει αποκρύψει μια απόδειξη 400 ευρώ και ένα άλλο έχει κλέψει εκατομμύρια, θα λέμε μόνο τα ονόματα και των δύο. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα ονόματα, αλλά και τα ποσά. Θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει ακριβώς για να πληρώνει ο κόσμος τους φόρους του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν. Νιούτον Ντανία, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω τον Ντόμ Νέιλεν. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι το 89 ιδρυθήκατε. Πριν από 23 χρόνια έχετε κάνει καμιά πρόοδο έκτοτε. Γιατί βλέπω τον τεράστιο ρυθμό φορολογικών παραδείσων που υπάρχουν ανά τη γη. Και εσείς και εγώ είμαστε από το ίδιο κράτος μέλλον. Έχει, δεν έχει καταργηθεί κανένας φορολογικός παράδεισος που προστατεύεται από τη Βρετανία και μάλιστα χρηματοδοτείται κιόλα. Εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Παρακαλώ με διορθώσετε αν κάνω λάθος και ελπίζω να ασφάλω. Και ένα δεύτερο ερώτημα είχα να σας κάνω. Είναι σωστό ο δικός σας οργανισμός να προτείνει πρότυπα για τα κράτη-μέλη. Στην Ένωση έχουμε 27 κράτη-μέλη και έχουν διαφορετικούς κανόνες, ποινές, κυρώσεις, νόμους, με τεράστια παραθυράκια και σε αριθμό. Δεν θα πρέπει να προτείνουμε να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τι νόημα έχει να έχουμε 187 πρότυπα παγκοσμίω πείτε μου ότι προτείνετε κάτι, μια εγκάρσια εναρμόνιση διεθνή, διορθώστε με. Και κάτι αντίστοιχο θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Μπάση. Εσείς στη δουλειά σας δεν θα πρέπει να προτείνετε εναρμονισμένους κανόνες για το σύνολο της Ένωσης. Εσείς μιλάτε για μεμονωμένα κράτη-μέλη. Εμείς θέλουμε ε, ευρωπαϊκούς κανόνες, νόμους, ποινές, τιμωρίες και σύστημα αποκάλυψης, όχι εθνικά συστήματα. Ευχαριστώ. Eh, Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στον εκπρόσωπο της ΦΙΕΤΙΦΗ θα ήθελα να ρωτήσω Πώς παρακολουθείτε στον οργανισμό σας το ρόλο που παίζουν ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διακίνηση και στην ανακύκλωση. Και αυτό λόγω της αδιαφάνειας και της ανεπάρκειας των εθνικών κανόνων και στην προκειμένη περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας με τη διατήρηση ιστορικών δομών όπως η City of London Corporation που φαίνεται να ανήκει σε άλλες εποχές, άλλες ιστορικές εποχές και φαίνεται τελικά να εκπροσωπούν ένα κράτος εν κράτη. Ποιες είναι οι πραγματικές εξουσίες έναντι αυτών των φορολογικών παραδείσων μεταξύ αυτών και μία από τις ε, χώρες ιδρυτές της Ένωσης, το Λουξεμβούργο. Πώς μπορείτε εσείς λοιπόν να παρεμβαίνετε και να βρίσκετε όλα τα μυστικά. Δείτε τι έγινε στην περίπτωση Μαντόφ. 55 δισεκατομμύρια δολάρια επενδυμένα από κόσμο ο οποίος ε, πίστηκε διότι οι επιχειρήσεις του Μαντόφ έδρευαν στο Λουξεμβούργο που θεωρείται μια πολύ σοβαρή και αξιόπιστη χρηματοπιστωτική αγορά και είναι και μία χώρα ιδρύτρια. Αυτά για τον FATF. Πώς μπορείτε εσείς να έχετε νέα, να έχετε πληροφορίες όταν το Λουξεμβούργο δεν επιτρέπει σε εισαγγελείς από τρίτες χώρες που κάνουν έρευνες για ε, χρηματοπιστωτικά εγκλήματα, δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση. Τώρα για τον, προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Φυσικά μήπως θα ήθελε να μας πει κάτι και αυτός. Εγώ για το ρόλο της ε, City θα ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο στις 27 Αυγούστου του 10 ανέφερε η Daily Express. Το έλεγε ένα, ο επικεφαλής ε, της ε, ε, Σοβιετικής Εισαγγελίας που έλεγε ότι το Λονδίνο είναι το στεγνοκαθαριστήριο του άπλητου χρήματος. Δείτε τι λένε δηλαδή σοβαροί άνθρωποι. Είναι, και τελικά σε αυτό το πλυντήριο συχνάζουν πολλά, πολύ ισχυροί πελάτες. Μπορούμε, μπορεί να γίνει λοιπόν μία αναφορά για τις συγκεκριμένες δυσκολίες και για το πώς κανείς μπορεί να αντιδράσει έναντι αυτών των νομικών θεσμικών ε, σχημάτων γύρω από, την, ε, ε, γύρω από το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Διότι τελικά εμείς είναι σαν να θέλουμε να αποφύγουμε τις πλημμύρες ε, χωρίς ε, να καθαρίζουμε τα αυλάκια της αποχέτευσης. Παρακαλώ συντομεύετε λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι το παγκόσμιο δίκτυο των, παρα... των φορολογικών παραδείσων τα μεταφέρουν στις ε, διάφορες αγορές offshore μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσιο, να ρωτήσω κι εγώ. Να ρωτήσω κάτι όμως κατευθείαν, χωρίς ε, πολλές ζυριτζάντζουλες. Οι συνάδελφοι ανέφεραν τις τράπεζες ε, και το ρόλο τους στην ανακύκλωση. Φαίνεται πολλές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους κώδικες τους ε, δεν έχουν συμπεριλάβει την αυτοανακύκλωση. Εδώ και μερικά χρόνια γίνονται απόπειρες ε, για διεθνείς έρευνες στο Βατικάνο, στο Βατικανό, για την τράπεζα του Βατικανού, την ΙΟΡ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Δίνω το λόγο στον Τόμ Νίλεν και μετά ο Γκομπάση. Um, Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Αρχίζοντας με τη δική σας ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Το Βατικανό και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα, πράγμα το οποίο ε, συνέβη μετά από τις δραστηριότητες που ανακαλύφθηκαν από την ειδητή και ομάδα της Τράπεζα της Ιταλίας που ασχολείται με αυτά τα θέματα και τις ε, έρευνες που έπρεπε να γίνουν. Βεβαίως είναι εκτός των δραστηριοτήτων της ΦΙΑΙΤ και δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε τίποτα. Εμείς όμως πρέπει να πω ότι αναφέραμε το γεγονός στο αντίστοιχο φορέα του Συμβουλίου της Ευρώπης που έκανε μία αξιολόγηση του Βατικινού, συζητήθηκε τον Ιούνιο και εγκρίθηκε τα αποτελέσματα ώστε να μπορέσουν να κάνουν ε, μελέτη και αναθεώρηση των προβλημάτων που εμπίπτουν στα πλαίσια της δικής τους αρμοδιότητας. Και έτσι και νομίζω ότι υπάρχει βελτίωση. Τώρα, και από το ίδιο το Βατικανό υπάρχουν κάποια μέτρα, αλλά δεν μπορώ να σα πω μέχρι ποιο σημείο έχουν προχωρήσει. Τώρα, για να ασχοληθώ σύντομα με άλλε ερωτήσει. και όχι απαραίτητα με την σειρά με την οποία ζητήθηκαν, αλλά με μια λογική σειρά. Μια ερώτηση από τον κύριο Νιούτον Ντάν για το εάν ή γιατί δεν έχουμε ένα αρμονισμένο σύστημα που να εφαρμόζεται σφαιρικά παρά να έχουμε ένα σύστημα προτύπων και κανόνων που να ερμηνεύονται διαφορετικά σε κάθε χώρα. Η απάντηση είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συνάδει με την ε, φύση του οργάνου. Πρέπει να έχουμε συστήματα και κανόνες που να εφαρμόζονται από τον καθένα. Εδώ έχουμε ένα σύνολο ε, συστάσεων και ερμηνευτικές διατάξεις σχετικά με αυτό που κάνουμε και δίνουμε σε μεγάλες λεπτομέρειες ότι περιμένουμε από κάθε χώρα να κάνει στον τομέα αυτό. Πρόκειται λοιπόν για θέματα τα οποία είναι τεχνικά και δίδουμε εμείς την κατάλληλη αξιολόγηση λεπτομέρως. Εδώ Φερρυπίν σε 150 σελίδες έκθεση αναφέρουμε για την Ισπανία όλα τα μέτρα τα οποία έλαβε η χώρα αυτή για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα, την ε, νομοθεσία, τις τεχνικές αδυναμίες κτλ. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται στα πλαίσια κάθε εθνικού νομοθετικού συστήματος, αλλά ως φορέας εμείς Θέλουμε να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον μια εναρμονισμένη προσέγγιση και να μπορέσουμε όλα αυτά να μεταφέρουμε στην ε, κοινοτική νομοθεσία είναι πραγματικό εφιάλτης και χαιρόμαστε που η Κομισιόν παίρνει κάποια μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση επίσης. Τώρα κάποια ε, ερωτήματα τέθηκαν για θέματα ε, φορολογικά. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα πάντα για να καταπολεμήσουμε το ε, οικονομικό έγκλημα. Έχουμε στα πλαίσια της δουλειά μας αναλάβει και αυτό το θέμα που εφέτος το Φεβρουάριο και το προσθέτουμε στην σειρά μέτρων πρέπει να λάβουμε για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις ε, οικονομικές παράνομες δραστηριότητες. Βεβαίως είμαστε και στενοί στην εργασία με τον ΩΣΑ για την ε, ανταλλαγή απόψεων πληροφοριών και να εναρμοστούμε σε αυτό το οποίο γίνεται και σε εκείνο το επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι ένα από τα κύρια όργανα που υπάρχουν ε, είναι η Financial Intelligence Unit, η υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος που υπάρχει σε όλες τις χώρες και εμείς θέλουμε να έχουμε πληροφορίες και λαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Τώρα, αν όλα αυτά δεν δίδονται απευθείας στις ε, ομάδες δίωξης αυτές, είναι διότι πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ βέστες σε παραλαμβάνω. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε εμείς όλα αυτά τα στοιχεία να τα εξετάσουμε με ασφάλεια και να μην τύχουν ε, τις εξέτασεις που γίνεται συνήθως σε ε, οικονομικές προβλήσεις, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ε, όλα αυτά τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Και βεβαίως θέλουμε πάντα να γίνονται σε τις προφορίες τις οποίες χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούν οι άλλοι. Τώρα, όσον αφορά το ξέπλυνα, ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τα πρόστιμα πρέπει να, να επιβάλλονται σε διάφορες τράπεζες. Οι κυρώσεις, εάν κανείς δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσει δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι οι τράπεζες ιδιαίτερα προσεκτικές ώστε να εντοπίζουν τέτοιου είδους οικονομικές δραστηριότητες, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι αν μια χώρα δεν μπορεί να επιβάλλει τέτοιου είδους κυρώσεις και αν ε, η συμπεριφορά κάποιων ε, τραπεζών δεν είναι κατάλληλη και δεν ε, λαμβάνεται ιδέους επιμέλεια εκ μέρους τους ώστε να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις είναι κάτι το οποίο εμείς το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάση το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι επιτρέψτε μου αρχίζοντας να πω στον κύριο Νιούτον Τάν ότι αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να εισαγαγούμε είναι ένα γενικότερο κοινοτικό πλαίσιο, ένα σύνολο κοινοτικών κανόνων. Δεν λέω βεβαίως ότι θα πρόκειται για μία εναρμόνιση σε ανατοτόριο, θα πρόκειται για μία οδηγία και θα πρέπει να μπορούν να γίνονται οι διάφορες προσαρμογές ανάλογα με την κάθε εθνική συζήτηση. Αλλά σε γενικότερα πλαίσια θα πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βοήθεια πραγματικών κοινοτικών, ευρωπαϊκών κανόνων. Τώρα, όσον αφορά στην προσέγγιση που βασίζεται στο ρίσκο. Και πάλι θα πρέπει να πω το εξή στον εισηγητή. Αυτό που έχουμε κατά νου δεν είναι να μειώσουμε τις εξουσίες που διαθέτουν σήμερα, αλλά να τις αυξήσουμε αντιθέτως. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, οι κανόνες μας δεν θα είναι αυστηροί. Το αντίθετο. Θέλουμε όμω να έχουμε ένα μηχανισμό που να βασίζεται σε αποδείξει και σε μαρτυρίες και σε όλα τα κράτη-μέλη και όλα τα άτομα και βερίς που θα καλύπτονται από την οδηγία θα πρέπει να καταλαβαίνουν, να κατανοούν τους κινδύνους που έχουν στους τομείς του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και σε περιπτώσεις διαφορές. Γι' αυτό οι κανόνες θα πρέπει να είναι διαφανείς και να είναι και από τις εθνικές εποπτικές αρχές και βάσει αυτής της αξιολόγησης θα μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως λιγότερη δέουσα επιμέλεια όταν αυτό δικαιολογείται, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας όταν υπάρχει κίνδυνος εμφανός. Λοιπόν, τα πράγματα θα γίνονται με λιγότερο αυτόματο τρόπο, αλλά περισσότερο ε, βασιζόμενο στην πραγματική κατάσταση. Ο στόχος λοιπόν είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ισχυρούς τους κανόνες, παρά πιο χαλαρούς. Τώρα, όσον αφορά τα φορολογικές παράνομες πράξεις και εγκλήματα, βεβαίως θα βοηθηθούν οι πάντες και θα είναι πιο εύκολη η ζωή όλων μας εάν μπορέσουμε να εναρμονίσουμε την πολιτική μας όσον αφορά τα ε, προβλήματα αυτών των μεταφορικών. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι στο ευρωπαϊκό σύστημα όταν μιλούμε για τέτοιου ε, είδους ε, ε, φορολογική εναρμόνιση θα πρέπει να έχουμε ομοφωνία από το Συμβούλιο και όπως λένε και οι Γάλλοι το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Λοιπόν, ή θα κάνουμε κάτι το αποτελεσματικό και χρήσιμο στον τομέα αυτό του ε, ξεπλήματος παράνομου χρήματος ή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πλήρη εναρμόνιση, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε επίπεδο Συμβουλίου για να επιτύχουμε την ομοφωνία για τους λόγους που κάποιοι από εσά αναφέρετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα απευθυνθούμε και αυτό το, δεν, θα, δεν θα ασχοληθούμε και με το θέμα των φορολογικών παραδείσεων. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι, συγγνώμη κανένα, εξετάζουμε το θέμα αυτό εκ του και μαζί με τον συνάδελφο σε μέτα που είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά της φορολογικής πολιτικής προσπαθούμε να δούμε πώς θα απευθυνθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό των φορολογικών παραδείσων. Αυτό όμως γίνεται εκ παραλίλου και δεν θα πρέπει να το συγχαίουμε με αυτά τα οποία θα κάνουμε εμείς στα πλαίσια της νέας πρότασης που θα υποβέλουμε, διότι διαφορετικά το μόνο αποτέλεσμα θα είναι ότι η έγκριση της πρότασης που θα σας προτείνουμε σύντομα θα αναβάλλεται ΕΣΑΗ και δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Αποφάσισα να καλύψω τα κύρια θέματα που τέθηκαν, ίσως ε, όχι με τη σειρά, αλλά αν θέλει κάποιο μια συμπληρωματική απάντηση, ας μου το πει, με στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ. Τελειώνουμε με αυτό το πρώτο πάνελ. Σας ευχαριστούμε για όσα μας και ε, όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σίγουρα θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων. περαιτέρω και για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όσα είπατε στην τελική έκθεση, σας παρακαλώ να μας δώσετε ένα έγγραφο με τις τοποθετήσεις σας. Allora, noi adesso passiamo... Πάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. κανάλια και τεχνικές ανακύκλωσης του χρήματος και μέσα και τεχνικές ε, για τη διαπίστωση και την καταπολέμηση. Θα ακούσουμε τον Σαν Κλοντ ε, που είναι πρόεδρος της, ε, μονάδα, της μονάδας κατά της ανακύκλωσης του Βελγίου. Μετά τον Αντώνιο Μαρία Κώστα, ο οποίος είναι γενικός αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και θα μιλήσει για το ξέπλυμα του χρήματος που προέρχεται από το ναρκωτικά. Ο Ίγκο Φίντλερ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από το παράνομο παιχνίδι, από τον τζόγο. Και μετά ο Ρενεουάκ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των κινδύνων στο τραπεζικό τομέα. Δέκα λεπτά ο καθένας εισηγητής και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. με τον εισηγητή και τους συντονιστές. Ο Ζαν έχει το λόγο, 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με έναν τρόπο σχετικά παράδοξο. Θα σας θυμίσω μερικά νομοθετικά κείμενα τα οποία αναφέρθηκαν, τις ε, συστάσεις του ΦΙΕΤΙΦΗ, όλες τις ε, κοινοτικές οδηγίες και αυτό δεν το κάνω εδώ απλά και μόνο για να σας τα υπενθυμίσω όλα αυτά. Απλώς ε, θέλω να σας αναφέρω ότι, μέσα, ότι σε όλες αυτές τις πτυχές υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο εκπροσωπώ εγώ, είμαι ένας άνθρωπος ε, που εργάζομαι επί τόπου. Και λέγω, θα σας πω ότι υπάρχει ο κανόνας αλλά και η εφαρμογή του κανόνα. Αυτό θα σας έλεγαν και άλλοι συναδελφοί μου από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Εμείς ε, στο Βέλγιο εφαρμόσαμε όχι μόνο τις συστάσεις του Φιλίππη, αλλά και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τις εφαρμόζουμε εδώ και 20 χρόνια. Από τις 11 Ιανουαρίου του 1993. Και πρόκειται για ένα νόμο που θέλει να προλάβει την ανακύκλωση του βρώμικου χρήματος και το ξέπλυμά του, αλλά και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η Financial Intelligence Unit, η FIU, στο Βέλγιο, η Μονάδα Χρήματο-Οικονομικών Πληροφοριών κλπ. Είναι μια λειτουργική μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα και είμαστε και μια διοικητική ομάδα, μονάδα ταυτόχρονα. Στην ε, FEU έχουμε διάφορα, διάφορους, ε, διάφορα στελέχη, έχουμε διοικητικούς, ε, δικαστικούς και αστυνομικούς. Εγώ θέλω να σταματήσω μια φήμη που κυκλοφορεί πολύ συχνά και που λέει ότι αυτοί, αυτές οι μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι είναι ετερόκλητες. 20 ε, χρόνια κάνω εγώ αυτή τη δουλειά και πρέπει να σας πω ότι στις ΦΙΑΙΟΥ δεν αλλάζει ιδιαίτερα το ρόλο της, είτε είναι διοικητική, είτε είναι δικαστική, είτε είναι αστυνομική. Λειτουργούν κάλλιστα πολύ ωραία μεταξύ τους όλες αυτές οι μονάδες, με τις αστυνομικές μονάδες, με τις ε, δικαστικές μονάδες, με τις μονάδες πληροφοριών. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν δημιουργεί πραγματικά προβλήματα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς έχουμε δύο υπουργούς πάνω από τα κεφάλια μας. Τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί εμείς έχουμε και την οικονομική πλευρά υπό την αρμοδιότητά μας αλλά και την δικαστική πλευρά διότι το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος είναι μια εγκληματική δραστηριότητα η οποία αφορά και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και στο δικαστικό διότι χρειάζεται η καταστολή. Καταστολή κυρίως ε, υπό την έννοια ότι πρέπει να πάρουμε εμείς ε, αυτά τα λεφτά τα οποία έχουν ανακυκλωθεί και λευκανθεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα μεταξύ του νομοθετικού, της νομοθετικής και πρακτικής πλευράς. Υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχετε σαφώς κατά νου. Αυτό το σύστημα πρόληψης ε, βασίζεται σε ένα σύστημα συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί εδώ και 20 χρόνια. Καταρχήν με το ιδιωτικό ε, με τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα και μετά με τον ιδιωτικό μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι ένα risk-based approach. Εδώ και 20 χρόνια λειτουργεί αυτό το σύστημα. βάσει των αρχών της ΦΕΙΤΙΦΗ και λειτουργεί μια χαρά αυτό το σύστημα διότι υπευθυνοποιεί τους ε, αρμόδιους. Μπορούμε βεβαίως να εργαστούμε και πληροφοριοδότες ε, και επίσης προσπαθούμε να να συνεργαζόμαστε και στο επίπεδο των πληροφοριών, γι' αυτό θα σας τα πω αργότερα. Η διαπίστωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η διαπίστωση των κινδύνων, αλλά και το profiling. Και όταν λέω profiling, μιλάω για την ισορροπία του ιδιωτικού βίου και της διαδικασίας ε, ε, εξεπλήματος. Δεν είναι πάντα εύκολο να κάνει κανείς profiling για ε, κάποιο πελάτη ο οποίος ε, κάνει ορισμένες συναλλαγές όταν θέλουμε να σεβαστούμε όλες τις οδηγίες σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού βίου. Πρόκειται για κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει όμως να, να προσέξουμε αυτή η δύσκολη διαδικασία που πρέπει να παραμείνει ε, δύσκολη. Πρέπει να προσέξουμε αυτό το σύστημα να μην επιτρέψει στους αντιπάλους μας, δηλαδή τους εγκληματίες, να προχωρούν, να, κάνουν καταχρήσεις και να επεξεργάζονται στρατηγικές, ακόμη πιο μπερδεμένε και ε, δύσκολες να διαπιστωθούν. Γίνεται μία δήλωση υποψίων στην ε, μονάδα μας και βασίζεται είτε απλά σε υποψίες είτε σε γεγονότα. Τώρα η μονάδα του οικονομικών πληροφοριών αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των ε, δικαστικών αρχών και των αρχών που υποβάλλουν ε, την αναφορά. Μπορούμε δηλαδή εμείς ε, να ενημερώνουμε τις δικαστικές αρχές. Εμείς προστατεύουμε και αυτόν που δηλώνει και τον πελάτη όμως. Διότι όλα αυτά φυσικά καλύπτονται από μια ενισχυμένη μυστικότητα. Η διεθνή συνεργασία μεταξύ των ε, μονάδων οικονομικής πληροφόρησης. Εμείς έχουμε 80 συμφωνίες συνεργασίας. είναι 100% το, να πούμε ότι είναι 100% λειτουργικές όλες αυτές οι συμφωνίες ε, δεν θα ήταν ακριβές. Άλλες είναι πιο λειτουργικές από άλλες. Σε αυτόν τον τομέα όταν ψάχνουμε εμείς εγκλήματα, να ζητούμε εγκλήματα, έχουμε το τυπικό μέρος που αφορά στον ε, τυπικό σεβασμό των, ε, της νομοθεσίας Η μονάδα μας, η FIU, δεν πρόκειται να σταθεί όμως αυτό το τυπολογικό σχήμα, αλλά στην αποτελεσματικότητα. Εμείς προσπαθούμε πάντοτε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες πληροφορίες για αποτελεσματική, που οδηγούν και στην αποτελεσματική λειτουργία. Φυσικά έχουμε την αμοιβαιότητα, τη μυστικότητα και την ε, συμφωνία την εκ των προτέρων για την ε, δημοσιοποίηση πληροφοριών. Μετά έχουμε τις τυπολογικές αναλύσεις. Έχουμε όμως και τις στρατηγικές αναλύσεις που μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε περισσότερο μία προσέγγιση που βασίζεται σε ένα ρίσκο και σε μία απειλή που μπορούμε να τη διαπιστώσουμε είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε διεθνώς. Σας παραπέμπω στην ετήσια εκθεσή μας, βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Και ένα τελευταίο σημείο ε, σημαντικό, όπου μία μονάδα παίζει σημαντικό ρόλο, είναι η αξιολόγηση του κινδύνου για, την, για το ξέπλυμα των κεφαλαίων που αποτελεί και υποστήριξη για τον καθορισμό των στρατηγικών πολιτικών και την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλειών και επισήμων δράσεων. Μας είπαν μέχρι τώρα ότι το ΣΕΦΑΙ μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικό και συγκρατημένο στη δράση του. Εμείς έχουμε όμως στοιχεία. Το 2016 1.165 καταγγελίες έλαβε η υπηρεσία μας που αντίστοιχα φτιάξαμε τα, διάφορες, τα διάφορα ντοσιέ. 4.479 ντοσιέ και το συνολικό ποσό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως πρόκειται για τα ποσά τα οποία εμείς έχουμε απλώς διαπιστώσει. Δεν τα έχουμε κατάσχει, δεν έχουμε ακόμη καμία δικαστική απόφαση. Εδώ στο Βέλγιο έχουμε 2 δις ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το χρήμα έχει κερδιθεί εδώ στο Βέλγιο με εγκληματικές δραστηριότητες. Πρόκειται για ε, κινήσεις κεφαλαίων που τα διαπιστώνουμε να βρίσκονται στο Βέλγιο είτε και μπορεί να μην βρίσκονται ακόμη στην επικράτειά μας. Πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς ε, όταν μιλάμε για αυτά τα ποσά, αλλά νομίζω ότι ήδη το ποσό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το φαινόμενο. Τώρα πώς συμβάλλει ο καθένας. Βλέπετε ότι τα χρηματιστηριακά γραφεία και οι τράπεζες είναι αυτά που συμμετέχουν στο μεγαλύτερο βαθμό. Πρέπει να τονίσουμε όμως των αντίον ότι υπάρχουν και άλλοι εγκινδύνο τομείς, ε, άλλοι κλάδοι, διότι δεν συμμετέχουν επαρκώς στην καταπολέμηση του ξεπλήματος. Έχουμε ε, ε, ένα σωρό επαγγέλματα. Λογιστές, ελεγκτές ε, και άλλους κλάδους απόλυτα νόμιμους. Εμείς έχουμε έναν πίνακα εδώ. Έχετε εδώ τις διάφορες υποψίες που έχουμε λάβει. Βλέπετε τον αριθμό των όσων έκαναν την δήλωση. Ε, βλέπετε συνολικά ποιος είναι ο αριθμός των επαγγελματιών και πόσοι είναι οι υποπτοί. Και βλέπετε πόσο μικρό είναι το ποσοστό για το κάθε επάγγελμα. <coughs> Σας παρακαλώ δόκρετε. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα ε, για τον κίνδυνο, ε, ο οποίος ε, είναι ιδιαίτερα υποτιμημένος προς στιγμήν, κυρίως όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της απάντησης και στην ταχύτητα. Υπάρχει ένας κίνδυνος διείσδυσης αυτών των ποσών και πρέπει να γίνεται ανάλυση κινδύνων όχι μόνο των κινδύνων που αντιπροσωπεύουν για μας οι εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και τον κίνδυνο που και εμείς οι ίδιοι αντιπροσωπεύουμε ε, για, τον τρόπο που, που δρούμε. Έχουμε μία σημαντική δυσαναλογία μεταξύ των μέσων που διαθέτουμε και των ε, νομικών δυνατοτήτων που έχουμε και όλα αυτά είναι πάρα πολύ, είναι ελάχιστα απέναντι στην δύναμη των εγκληματικών οργανώσεων. Μετά μιλάμε εμείς για tax crime, για φόρο του εγκλήματος. Αλλά μέγα μέρος της αδιαφάνειας ε, οφείλεται στο φορολογικό σύστημα, διότι τελικά όλοι αυτοί εκμεταλλεύονται όλα τα παραθυράκια του φορολογικού συστήματος, διαφεύγουν κεφάλαια ε, στο, στους φορολογικούς παραδείσους. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα υπάρξει, υπάρχει και θα υπάρξει για πολύ καιρό. Επίσης υπάρχει και το θέμα των, ε, της κληροκεφαλιάς. Έχουμε πολλές φορές εμείς ιδέες απόλυτα ριζωμένες και το βλέπουμε αυτό για το πώς αντιδρούμε δηλαδή στην αντιμετώπιση και της τρομοκρατίας και των εγκληματικών οργανώσεων. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια, ένα ανοιχτό πνεύμα, μια ενορατικότητα ε, για την καταπολέμηση όλων αυτών των οργανώσεων. Προχωράμε πολύ αργά και αυτό το οποίο μας καθιστά ε, αποτελεσματικούς είναι η διαφορά αυτό το οποίο μπορεί απλώς να θεωρηθεί αποτελεσματικό είναι η διαφορά του, μεταξύ του ποσού το οποίο διακινείται και αυτού που πραγματικά πιάνουμε. Πρέπει λοιπόν εμείς να αυξήσουμε την δυνατότητα κράτησης αυτού του χρήματος, διαπίστωση και κράτηση του χρήματος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Jean-Claude ο Αντώνιο Μαρία Κώστα Κύριε Πρόεδρε, οι συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου συνήθως έχουν ως θέμα την ανάπτυξη, την ειρήνη, την ασφάλεια. Σήμερα είναι διαφορετική η συνεδριασή σας, διότι αφορά θέματα τα οποία δεν είναι ευγενή, αλλά αρνητικά. Δεν μιλούμε για παραγωγή, αλλά για καταστροφή. Δεν μιλούμε για εμπόριο, αλλά για εμπορία. Δεν μιλούμε για επενδύσεις, αλλά για ε, νημοποίηση εσόδων από εγκλήματα. Πρόκειται για την οικονομία του εγκλήματος, μια γιγαντιαία επιχείρηση μεγαλύτερη από το Fortune 500.000. Όλοι γνωρίζουμε πώς έχουν τα πράγματα στο παρελθόν και τα τελευταία 25 χρόνια. Το έγκλημα το οικονομικό έγινε οργανωμένο, διακρατικό, πήρε μία διάσταση μακροοικονομική και απορρέει ε, και ε, τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του τα παίρνει, τα αντλεί από την παγκοσμοποίηση. Έχει τα κοινοβούλια, στις κυβερνήσεις, κατέστρεψε χώρες, άλλαξε τις στρατηγικές επιχειρήσεις, διαφοροποιήθηκε και από τα ναρκωτικά, τα όπλα, ε, τους ε, φυσικούς πόρους, τα απόβλητα, πέρασε και σε άλλους τομείς όπως του κυβερναγκλήματος, της ε, τρομοκρατίας, η εγκληματίες του τομέα αυτού είναι οι πρώτοι οι οποίοι μετακινούνται όταν υπάρχουν ε, διάφορες ε, ευκαιρίες τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Πρέπει να πω ότι πριν από δέκα χρόνια όταν άρχισα να εργάζομαι στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και Οικονομική Οικονομικά, ε, ήμουν ο πρώτο ο οποίο έκανε την πρώτη έκθεση με τίτλο Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματο, το οποίο ήταν μια πραγματική πρόκληση. Και τότε μπορούσαμε να έχουμε έγγραφα τα οποία αφορούσαν τον ε, αγορά η οποία όλο και περισσότερο, την εγκληματική αυτό το τομέα, ο οποίο επεκτάθηκε όλο και περισσότερο ανά τον πλανήτη, όπου είχαμε να κάνουμε με παράνομα αγαθά, τα οποία προέρχονταν από μία ήπειρο και περνούσαν στις άλλε. Υπάρχει ένας ε, τομέας του εγκλήματο, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο καλύτερα κατανοητός από όλους. Πρόκειται για την παράνομη εμπορία ε, ελεγχόμενων ουσιών όπως το όπιο, ηρωίνη, κοκαίνη και διαγερτικές χημικές ουσίες όπως έκσταση και μαριχουάνα. Από την μεριά της προμήθειας ξέρουμε ότι σήμερα 850 τόνοι κοκαίνης προέρχονται από τις χώρες των άνθρωπων, 550 τόνοι ηρωίνης από το Αφγανιστάν, 600 τόνοι συνθετικών ε, ναρκωτικών ουσιών και 40.000 τόνοι κάναβης βρίσκονται στις παγκόσμιες αγορές. Οι χώρες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες παράγουν αυτές τις παράνομες ουσίες όπως το Αφγανιστάν με το όπιο και η Κολομία με την ε, ε, κοκαίνη είναι αυτές στις οποίες εστιάζεται η μεγαλύτερη προσοχή. η περισσότερα ωφέλη, τα κέρδη από τα ναρκωτικά ε, γίνονται κυρίως προς όφελος των πλουσίων χωρών. Παραδείγματο χάρη από την ε, ε, παγκόσμια αγορά των περίπου 55 δις για την ηρωίνη του Αφγανιστάν, μόνο 5%, 2,3 δις ε, πηγαίνουν στους αγρότες του Αφγανιστάν, στις ε, ομάδες εξεγερμένων και στους εμπόρους. Από τα 72 δις της κοκαίνης, το 70% των κερδών περνούν από τα χέρια των ε, μεσαζόντων στις χώρες που καταναλώνουν αυτά τα ναρκωτικά και 20% πηγαίνουν εκτός των, χωρών παραγωγής. Από την πλευρά τώρα της ζήτησης πρέπει να πω ότι περίπου 200 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν ναρκωτικά μια φορά το χρόνο, ενώ 25 εκατομμύρια ε, είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερο από 1% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι εθισμένο. Και θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το καπνός χρησιμοποιείται από το 1 τρίτο του πληθυσμού και η νοπνευματώσεις από 1 τέταρτο. Ετησίως πρέπει να πω ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν μισό εκατομμύριο άτομα παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν τρομερό αριθμό που βεβαίως αναλογικά είναι μικρότερος από τα άτομα τα οποία πεθαίνουν κάθε χρόνο ε, επειδή είναι καπνιστές ή καταναλώνουν υνοπνευματόδη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε να κάνουμε με απαγορευμένες ή με επιτεπτές ουσίες. Η Ευρώπη ε, είναι η μεγαλύτερη αγορά ηρωίνης, ενώ η Ρωσία η μεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης ανά τον κόσμο, 70 τόνοι. Η αγορά της κοκαίνης ε, στην ε, Βόρεια Αμερική, παρά το γεγονός ότι συρρυκνώνεται, παραμένει η μεγαλύτερη ανά τον κόσμο. Πράγμα το οποίο δημιούργησε ε, στο, πόλεμο των ναρκωτικών στη, στη σύνορα Αμερικής με το Μεξικό. Από την Λατινική Αμερική η κοκαίνη μεταφέρεται μέσω της Αφρικής στην Ευρώπη και κάποιες χώρες της Δυτικής Αφρικής κινδυνεύουν να καταστραφούν. Έχουμε να κάνουμε με την ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών που πολλές φορές στρεβλώνει ακόμη και τα ίδια τα οικονομικά θεμέλια της περιοχής, δημιουργεί υποανάπτυξη και προβλήματα στα τοπικά νομίσματα. Έχουν ε, ε ε, διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την απειλή από τα ναρκωτικά. Κάποιοι μιλούν και πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα υπεραπλουστευμένο μοντέλο για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά. Άλλοι επίσης με ε, πολύ απλουστευμένο τρόπο μιλούν για έναν κόσμο ελεύθερων ναρκωτικών, στον οποίο θα κυκλοφορούν ελεύθερα τα ναρκωτικά και μιλούν για νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Πρέπει να πω ότι αυτά τα δύο ελκυστικά επιχειρήματα είναι λανθασμένα. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι εδώ για να συζητήσω το θέμα του ελέγχου των ναρκωτικών, αλλά για να πω κάτι διαφορετικό. Ενώ η διεθνής κοινότητα γνωρίζει πως έχει κατάσταση με τα ναρκωτικά παγκοσμίω, πρέπει να πω ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι η πόσο για την σημαντικό είναι για την οικονομία αυτό το πρόβλημα και το πρόβλημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ακόμη δεν μπορέσαμε να ε, περιορίσουμε αυτούς τους στόχους και τον κίνδυνο που είναι για όλους της μαφίας και ξέρουμε ότι αυτό το οποίο ε, γίνεται είναι ότι οι εγκληματίες στον τομέα αυτό δεν έχουν πολιτική ατζέντα και ξέρουμε ποιο είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούν. Είναι εκεί για να μπορέσουν να ελαστοποιήσουν τους, ε, τους κινδύνους και να μεγιστοποιήσουν το όφελο χρησιμοποιώντας την διαφθορά. Ας δούμε πρώτα απ' όλα τον κίνδυνο. Πώς ενεργεί η μαφία. Προσπαθεί να δει που ενδεχομένως θα την ε, πιάσουν και αλλάζει η χώρα. Πηγαίνει εκεί που το κράτος δικαίου είναι ασθενές. Έτσι υπάρχουν δραστηριότητες παράνομες σε περιοχές σταθερότητας, σε περιοχές σύραξης και στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα ωφέλη, η απόδοση, κυρίως ε, η σχέση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και νομίμων δραστηριοτήτων. Η παγκόσμια μαφία δημιουργεί περί ωφέλη της τάξης των 300 δις ετησίων από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Πρόκειται για χρήματα τα οποία σήμερα μπαίνουν και στην νόμιμο τομέα της οικονομίας σε πάρα πολύ ε, ε, πλούσιες χώρες. Και τώρα φτάνω στο τρίτο θέμα που θέλω να δείξω, την διαφθορά. Τη στιγμή της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης βλέπουμε τη διείσδυση του χρήματος της μαφίας ε, στην, ε, στην τομέα της τράπεζας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ε, Στη δεκαετία του 60 όταν ε, οργανώθηκε παγκοσμίως η μαφία, τα χρήματά της κυκλοφορούσαν ανά τις χώρες σε ρευστό. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 70 η οικονομική ε, ενοποίηση της Ευρώπης και γενικότερα η άνθηση του διεθνούς εμπορίου οδήγησε τη μαφία στο να κάνει συναλλαγές μέσω ε, τραπεζικών πράξεων. Στη δεκαετία του 80 όλοι συνειδητοποίησαν τους κινδύνους που ε, ενέχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες και δημιούργησαν την ε, ΤΑΦΤ. Στην δεκαετία του 90 το γεγονό ότι θελήσαμε να κάνουμε πιο καθαρό τον τραπεζικό τομέα ε, λειτουργήσε σωστά. Και έτσι ξαναγύρισε η μαφία σε συναλλαγές σε ρευστό. Με έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσά τα οποία κατασχέθηκαν ανά τον κόσμο. Και σήμερα με την ε, οικονομική κρίση που διερχόμαστε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και κυρίως μετά από το, 2000, ε, από το 2008 δημιουργήθηκε πρόβλημα έλλειψης λεφτότητας στον οικονομικό τομέα και έτσι άρχισε να ε, διεισδύει και πάλι η μαφία στον τραπεζικό τομέα. Πρέπει να πω ότι παρόλα αυτά, κατά την άποψή μου, η εποπτεία έχει κατά κάποιο τρόπο ε, και ηθελημένα θα έλεγα δυστυχώς αποτύχει εκ μέρους των διοκτικών αρχών. Το 2010 είδαμε πώς δημιουργήθηκε αυτό το θεματικό πρόβλημα της ε, εταιρείας της ε, τράπεζας Βαχόβιας οι συνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε εδώ να κάνουμε με ανακύκλωση πολλών εκατοντάδων δις δολαρίων που προερχόταν από τα καρτέλ του Μεξικού. Και πολύ πρόσφατα η HCBC επίσης κατηγορήθηκε ότι ξεπλένει δισεκατομμύρια. Και το ίδιο έγινε και με άλλες τράπεζες, με την Citibank, με άλλες τράπεζες και δεν συνεχίζω. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία διεθνή τράπεζα η οποία δεν ενέχεται ενδεχομένω τέτοιου δραστηριότητε. Η δυνατότητα των διοκτικών αρχών να προσπαθήσει να αμβλύνει τι δραστηριότητε του οργανωμένου εγκλήματο, κατά την άποψή μου, εξαρτάται από την βούληση των κυβερνήσεων να ε, μπορέσουν με χειρουργικό τρόπο αυτή την μετάσταση της μαφίας στον τραπεζικό τομέα να την αφαιρέσουν. Αυτό ε, με κάνεις να πω αυτό που άκουσα τώρα τελευταία, ότι δεν ε, ψάχνει τις τράπεζες η μαφία για να ανακυκλώσει τα χρήματα. Οι τραπεζίτες είναι αυτοί που προσπαθούν να βρουν τα χρήματα της μαφίας. Σήμερα αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα αυτή την απειλή που έχει γίνει οργανωμένη, διακρατική, με διάσταση μακροοικονομική. Η ανταπόκριση που πρέπει να υπάρχει εκ μέρους όλων, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε αυτό το έγκλημα, πρέπει να βασίζεται στην ε, ε, δραστηριότητα την συγκεκριμένη εκ μέρους της κυρίως για να ταυτοποιήσει, να κατασχέσει και να επιβάλλει κυρώσους τους υπόψη τους. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε το οργανωμένο έγκλημα που είναι μια οικονομική δύναμη που ε, έχει και οικονομικά κίνητρα και προσδοκίες να μπορέσει να τιμωρηθεί. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να πω ε, απεσιόδοξα ότι υπάρχουν παραδείγματα ε, κατά διαφόρων τραπεζών οι οποίες ευρέθηκαν ένοχοι για ε, ξέπλυμα χρήματος και επιδείχθηκε εκ μέρους όλων έλλειψη βούλησης για να τιμωρηθούν. Ευχαριστώ. Ο Ίγκο λέει, από το Πανεπιστήμιο του ε, Αμβούργου για το, την ανακύκλωση του βρώμικου χρήματος και το τζόγο. Στο διαδίκτυο. Okay. So thank you very much for the invitation. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ε, θα μιλήσω για το ξέπλυμα χρήματος και τον Ιντερνετικό τζόγο. Ε, το ξέπλυμα χρήματος είναι η προϋπόθεση για το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο με τη σειρά του απειλεί την κοινωνία μας, την οργανωμένη. Είναι τεράστια μπίζνα όπως ακούσαμε αυτό το έγκλημα και ε, οι οργανωμένοι κλιματίες... Ε, Ε, είναι διεθνής. Ε, πάντα ε, εμείς προσπαθούμε να νομοθετήσουμε και αυτοί οι οποίοι είναι businessmen και επιχειρηματίες προσπαθούν και αυτοί να ξεφύγουν. Πρέπει λοιπόν τα έσοδα αυτά που έχουν να τα νομιμοποιήσουν. Έχουν κάποιες εγκληματικές δραστηριότητε. και έχουν βρει ένα καινούργιο τρόπο τώρα που είναι το ιντερνετικό στοίχημα ή ο τζόγος στο διαδίκτυο και είναι πραγματικά η κατεξοχήν μορφή εξεπλήματος. Είναι τεράστιες οι ροές ε, ε, μετρητών και η κυκλοφορία, δεν υπάρχει φυσικό προϊόν, μπορεί να κρυφθεί το ξέπλυμα και η νομιμοποίηση ε, χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται καμία φυσική παρουσία. Και πολλές φορές είναι και αφορολόγητα τα κέρδη από τα παίγνια. Όχι παντού, στη Γερμανία τουλάχιστον ισχύει αυτό που είναι η πατρίδα μου και ακούτε και από την προφορά μου στα αγγλικά ότι είμαι Γερμανός, ε, είναι αφορολόγητα λοιπόν τα έσοδα και αυτό είναι ενισχυτικό. Λοιπόν, είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στον τζόγο. Παράνομος τζόγος από μόνος του, που είναι μια παράνομη δραστηριότητα, ε, και ε, ταυτόχρονα είναι και αξιόπινη πράξη και κακούργημα. Βέβαια αυτό δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι σημαντικές. Οι παράνομες συναλλαγές που έχουν συμβεί προηγουμένως. Δηλαδή είναι προϊόν εγκλήματος το χρήμα που χρησιμοποιείται ε, για να πληρώσει κανείς ένα έσοδο από στοίχημα ή από παίγνια και ε, μπορεί να έρθει σε ένα νόμιμο λογαριασμό. Αυτό ίσχυε πριν. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, το τυχερό παιχνίδι και ε, ένας, ως ένας τρόπος για να πληρωθεί μια τέτοια παράνομη δραστηριότητα και αυτή είναι η τρίτη περίπτωση. Ε, θα σας δώσω τρία παραδείγματα για το πώς γίνεται αυτό. Και γιατί είναι τόσο εύκολο και τόσο φτηνό ταυτόχρονα ε, να χρησιμοποιούν τον Ιντερνετικό τζόγο οι εγκληματίες για να ξεπλένουν τα χρήματά τους. Λοιπόν, ας υποθέσουμε τώρα εδώ ότι είμαστε ένας πανέξυπνος και παμπώνιος εγκληματίας και θέλουμε να ξεπλύνουμε 10.000 ευρώ ε, παράνομα και να καταλήξουν στον νόμιμο λογαριασμό μας στην τράπεζα. Τι θα κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε μία κάρτα που έχουμε πληρώσει εκ των προτέρων, prepaid, Ας πούμε έχουμε πουλήσει λίγη κοκαίνη και ε, αγοράζουμε μια κάρτα που λέγεται Pay Safe Card, προπληρωμένη και πηγαίνουμε με αυτή την κάρτα να παίξουμε πόκερ ή σε ένα καζίνο ή σε ένα στοίχημα αθλητικό, στο τζόγο και πληρώνουμε. Και λέμε παίζουμε λοιπόν, βέβαια κάτι πρέπει να παίξεις, αλλιώς δεν μπορείς να εισπράξεις. Οπότε παίρνει και ένα μικρό μερίδιο ο διαχειριστής του παιχνιού που είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό γιατί τα κέρδη είναι πολύ ψηλά, η αναδιανομή είναι πολύ ψηλή, είναι ηλεκτρονικό το παιχνίδι και το προϊόν αφορολόγητο γιατί πολλές φορές ε, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση στα τυχερά παίγνια στο διαδίκτυο. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε τέτοιες ε, ρυθμίσεις, αλλά είναι πολύ μικρές. Αν δείτε το συνολικό μερίδιο της αγοράς τζόγου στο διαδίκτυο, είναι κυρίως ανεξέλεγκτος. Παράδειγμα, στη Γερμανία είναι τελείως παράνομο να παίζει κανείς πόκερ επιγραμμικά, δηλαδή στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά είναι η μεγαλύτερη αγορά online πόκερ η Γερμανία. Έχουμε και άλλες χώρες που είναι νόμιμη ε, η μορφή αυτή τυχερών παιχνιδιών. Εν πάση περιπτώσει ε, είναι εξέλεκτη αυτή αγορά. Πας λοιπόν εκεί και παίζεις και ε, σου μένουν 9.950 ευρώ και τα στέλνεις στο λογαριασμό σου και την ώρα που παίζεις ο διαχειριστής του προγράμματος δεν διώκεται ούτε καν φυσικά. Και ό,τι συμβεί μέχρι τώρα δεν ε, ε, εμπίπτει στον έλεγχο της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών, γιατί είναι στην ομίχλη. Ε, όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα θολό τοπίο. Ε, δεν ε, ανταλλάσσουν και πληροφορίες αυτοί που έχουν τέτοιες παροχές στο διαδίκτυο με ε, τους διώκτες οικονομικού εγκλήματος. Λοιπόν, από το πόκερ πηγαίνουν τα λεφτά σας στον τραπεζικό λογαριασμό κατευθείαν. Όπως σας είπα, δεν είναι τίποτα το ξεχωριστό αυτό ε, στη Γερμανία έχουμε την παριθμόν ένα αγορά. αυτή είναι μια μικρή περίπτωση των 10.000. Να το χοντρίνουμε λίγο το παιχνίδι. Είστε ένας μεσαίος dealer και έχετε 200.000 ευρώ, περίπου έτσι θέλετε να επενδύσετε, να αλλάξετε χώρα για να πάτε σε μια τράπεζα offshore ε, που δεν έχει ε, συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών με τη δικιά σας ε, χώρα και την μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών και θέλετε να κάνετε εκεί κατάθεση. Λοιπόν, και πάλι θα κάνετε ένα στοίχημα, θα χάσετε λίγα λεφτά βέβαια, 95% είπαμε είναι το ποσοστό πληρωμής και μετά τηλεφωνείτε στην τράπεζά σας και λέτε «Α, κέρδισα το jackpot στο λότο, στο διαδίκτυο, τεράστια λεφτά και θα σας δώσω και προμήθεια, έχω να επενδύσω, δώστε μου προϊόντα. Και σας προτείνει η τράπεζά σας ολόχαρη διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και τι έγινε, 200.000 λοιπόν μέτρητά που είχατε παράνομα έσοδα, ε, τα ε, ξεπλένετε. Γιατί δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν προέρχονται από παίγνια και από κέρδη στο διαδίκτυο. Τώρα, έρχομαι στο τρίτο παράδειγμα. Είστε ένας τεράστιος έμπορος ναρκωτικών και έχετε 200 εκατομμύρια τώρα. Τι κάνετε. Θα ιδρύσετε ένα καζίνο online. Έχετε σε ένα φορολογικό παράδεισο ε, χρήματα, λογαριασμό, ε, ρευστοποιείται και δημιουργείται ένα καζίνο, ψεύδο καζίνο, ε, με ε, κουλοχέριδες, εικονικούς, μπίνγκο, τόμπολες, δεν ξέρω τι και λέτε κοίταξτε πόσος κόσμος παίζει στο καζίνο μου και χάνει τα λεφτά του. Υπάρχουν χώρες που αυτό είναι νόμιμο ε, και εκεί πληρώνεται και φόρο και κάποιες άλλες δαπάνες. Μπορεί να είναι νησί αυτή η χώρα και θα χαρεί πολύ αν της δώσετε 10 εκατομμύρια σε δαπάνες και φόρους και τα υπόλοιπα είναι τελείως νόμιμα έσοδα τελικά και κέρδη. Γιατί ε, έχετε ένα καζίνο, είναι επιχείρηση και τα κέρδη είναι από το καζίνο. Και μετά στέλνετε το ένταλμά ε, το έμβασμά σας ε, όπως είναι στη Γερμανία. Τώρα, τι γίνεται με το, το ηλεκτρονικό cash, οι χρηματικές ροές. Ξέρετε πώς παίζετε, έχετε ένα λογαριασμό, έχετε έναν πάροχο που μπορείτε να παίξετε εκεί και μπορείτε να αποσύρετε και τα χρήματά σας μετά. Τώρα στις λεπτομέρειες αυτό πώς γίνεται. Έχουμε 235 διαφορετικές μεθόδους πληρωμών, αρχής γενομένης από ε, τις ε, πιστοτικές κάρτες. Στο τέλος κάτω-κάτω έχουμε τα μετρητά ε, με ενδιάμεσες δυνατότητες και 2.910 μορφές διαχειριστών, παρόχων και είναι μια δραστηριότητα, μια επιχείρηση που ε, και μια δραστηριότητα που κινείται με ταχύτητα τους ρυθμούς, πολύ μικρές εταιρείες ανά τον κόσμο, ξεφυτρώνουν από εδώ και από εκεί, χάνονται, εξαφανίζονται, κλείνουν. Ε, αυτή η τυχερών παιχνίων ε, κατανέμουν βέβαια τον κίνδυνό τους, το σπάνε και έχουν διάφορες μορφές ε, παιχνιδιών και μορφών πληρωμών. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί, δεν κάνουν πολύ μεγάλη διαφήμιση. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν ουσιαστικά τελικά. Ε, το βλέπετε στη διαφάνεια που σας δείχνω εδώ πόσο περίπλοκο μπορεί να γίνει ε, με τις διάφορες μορφές πληρωμών και πώς πηγαίνουν έρχονται τα χρήματα. Τελικά δεν ξέρετε ε, ποιος κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο και ποιος πληρώνει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να ανοιχνευθεί και το ξέπλυμα χρήματος τελικά ε, στο Ιντερνετικό παίγνιο. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ότι είναι χαμηλό το κόστος και χαμηλός ο κίνδυνος ε, ανείχνευσης, ε, ταυτοποίησης. Και είναι πιο φτηνό τελικά να νομιμοποιήσεις έσοδα ε, άρα αποφέρει περισσότερο το έγκλημα, άρα έχουμε περισσότερο έγκλημα. Γιατί είπαμε ότι είναι και λογικοί άνθρωποι οι οργανωμένοι εγκληματίες, δρούν με ορθολογικό τρόπο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, να μην είναι αφορολόγητα τα κέρδη. Γι' αυτό είναι τόσο φτηνή αυτή η επιχείρηση. Δεύτερον, ε, είναι δύσκολο να ανοιχνευτεί. Μπορεί όμως να ανοιχνευτεί. Το πρόβλημα είναι όταν είναι αγορές ανεξέλεγκτες και αρρύθμιστες. Χρειαζόμαστε ε, μια μορφή επιβολής του νόμου και επάταξης της παράνομης δραστηριότητας παιγνίων στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε ε, όλες τις μορφές παιγνίων στο διαδίκτυο και ως διαμαγείας να χαθεί η παράνομη δραστηριότητα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει καθόλου αρρύθμιστη αγορά και ανεξέλεκτη. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής που είναι ο πρόεδρος ομάδας εργασίας Έμπιτς και είναι ο κύριος Ρανεβάτη. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να παρουσιαστώ. Είμαι πρόεδρος της ομάδας εργασίας της EBIT, European Banking Industry Committee, αλλά ήμουν μέλος της στην ομίας στην Γαλλία που ασχολείται με την μεγάλη εγκληματικότητα και ήμουν υπεύθυνο για θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας και έχω λοιπόν ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τι διοκτικέ αρχές και τις τραπεζικέ αρχές. Αυτά για να καταλάβετε ακριβώ τι θα σας εκθέσω σήμερα. Οι τράπεζες έπαιξαν πρωτοποριακό ρόλο στην καταπολέμηση των ε, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες εδώ και 25 χρόνια περίπου. Ήμουν ένας από τους εκπροσώπους της Γαλλίας της ΓΑΦΗ όταν συντάξαμε τις πρώτες 40 συστάσεις με στόχο να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Οι πρώτες συστάσεις του Γκάφου αφορούσαν πρώτα απ' όλα την παράνομα έσοδα από, τη, από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Μετά ασχοληθήκαμε με το οργανωμένο έγκλημα, μετά την 11η Σεπτεμβρίου ε, ασχοληθήκαμε με τα θέματα της χρηματοδότησης της δημοκρατίας και σήμερα ασχολούμεθα με φοροδιαφυγή και τα θέματα των ε, εσόδων από το όπλο μαζικής καταστροφής. Πρέπει να πω ότι διευρύνθηκε λοιπόν ο τομέας ε, επαγρύπνησης για τέτοιες δραστηριότητες εκ μέρους όλων των τραπεζών, διότι από τη στιγμή από την οποία προσπαθεί κάποιο να φοροδιαφύγει μπορεί να είναι εν δυνάμει Θα έλεγα λοιπόν ότι αυξήθηκε το πεδίο επαγρύπνηση μας. Δεύτερον, αυτή η υποχρέωση τι σημαίνει. Ότι από αντικειμενική συνεργασία κατά του οργανωμένου εγκλήματος περάσαμε σε επαγρύπνηση περισσότερο ε, όλων των δραστηριοτήτων των τραπεζών και σε μεγαλύτερη συνεργασία. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες από την περίοδο αυτή και μετά έθεσαν μηχανισμούς σε κίνηση και σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο μέσων και διαδικασιών για ένα μη ευκατακρόνητο κόστος ενημερωτικά θα πω, αλλά είναι ο μόνος αριθμός που γνωρίζουμε ότι οι γερμανικές τράπεζες το 2006 εξέτασαν το κόστος της πρόληψης του ε, ξεπλήματος χρήματος τράπεζας και έφτασαν σε 770 εκατομμύρια ευρώ κόστος για να αποφευθεί αυτό το κόστος. Μόνον για τις γερμανικές τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η μελέτη αυτή είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ. Ε, ε, έκαναν λοιπόν σημαντικές προσπάθειες για να αποκτήσουν τα κατάλληλα μέσα οι τράπεζες. Θα σας πω ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, τι συστήματα πρέπει να θέσουν σε κίνηση. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες πρέπει να σας πω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο προβλήματα, δύο υφάλους. Πρώτα απ' όλα, δύο δυσκολίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υπέρ της μάξιμο ενοποίησης. Αν είχαμε ε, να επιλέξουμε μεταξύ κανονισμού και οδηγίας, τα περισσότεροι θα επέλεγαν τους κανονισμούς παρά να έχουν μία κατώτατο επίπεδο οδηγίες που για τους τραπεζικούς ομίλους σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες γιατί μία χώρα στην άλλη θα πρέπει να θεσπιστούν διαφορετικοί μηχανισμοί που να προσαρμόζονται στην κάθε τοπική ε, κατάσταση. Δεύτερη παρατήρηση, δεύτερη δυσκολία. Υπάρχουν άτομα τα οποία ανέφεραν τις κυρώσεις των τραπεζών λέγοντας ότι πραγματικά πολλές τράπεζες ε, από, τους, ε, Αμερικαν... από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές υπέστησαν κάποιες κυρώσεις. Διαπιστώνουμε ότι οι δραστηριότητες αποτροπής για την τρομοκρατία και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι μία δραστηριότητα με μηδέν ανεκτικότητα εάν δεν γίνουν ε, δηλαδή σεβαστοί οι κανόνες, οι κυρώσεις είναι άμεσα εκτελεστές. Και τελειώνοντας, για να τελειώσω την εισαγωγική μου παρατήρηση, πρέπει να πω ότι από το 1990 έχουμε να κάνουμε μεταφορά εξουσίας και υποχρεώσεων εκ μέρους των κρατών προς τον τομέα των τραπεζιών. Έχουμε ε, φοροδιαφυγή, φοροαπάτες, τρομοκρατικές δραστηριότητες, ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματος και τα, για να διαχειριστούν τα προβλήματα αυτά οι χώρες φαίνονται αδύναμες. Όλα αυτά μεταφέρονται στο τραπεζικό τομέα. Πρόκειται για πρόκληση, έτσι. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές υποχρέωσεις για τις τράπεζες. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι η σφαιρική προσέγγιση, και αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, είναι η προσέρμηση από το ρίσκο. Αυτό προέρχεται από το γεγονό ότι διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογή των τραπεζών από τη στιγμή από την οποία όλου μα ενδιαφέρει το ξέπλυμα του χρήματος, εάν δεν έχουμε την προσέγγιση μέσω ρίσκου, δεν θα ξέρουμε από πού να αρχίσουμε, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τώρα για να επανέλθω στις υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα, η γνώση του πελάτη. Αυτό είναι πρωταρχική σημασία. Και όταν μπήκα στο τραπεζικό τομέα, ε, με εξέπληξε ότι ζητούσαμε από του τραπεζίτε να ξέρει τον πελάτη του. Αν δεν ξέρει τον πελάτη σου και σε τράπεζα, πώ μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Θα δείτε όμω ότι αυτή η γενική αρχή τέθηκε σε εφαρμογή, αλλά δεν είναι προφανή. Γνώση του πελίτη. σημαίνει του, του πελάτη. Θα πρέπει να τον εντοπίσει, να το ξέρει κανείς. Αν είναι κάτι το προφανές για τον κάθε ιδιωτικό ε, πελάτη, στον οποίο ζητά κανείς την ταυτότητα, όταν έχουμε να κάνουμε με νομικά πρόσωπα ή με επιχειρήσεις είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος ε, που έχει τη νομική προσωπικότητα με την οποία έχουμε σχέση και που θα ανοίξει λογαριασμό. Και σε πολλές χώρες οι δημόσιες αρχές δεν μας βοηθούν και πολύ, δεδομένου ότι τα υποχρεωτικά μητρά στον οποία θα πρέπει να καταγράφονται οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν υπάρχουν. Άρα λέγουν ε, κάποιοι ότι θα πρέπει να ζητήσουν τα στοιχεία και να ταυτοποιήσουν το πελάτη οι τράπεζες. Θα κάνω έκκληση για αυτό το θέμα στα συμπεράσματά μου. Οι υποχρεώσεις λοιπόν των τραπεζών είναι περισσότερες και πιο δύσκολες όταν έχουμε να κάνουμε με ε, πελάτες υψηλού κινδύνου, όταν έχουμε πολιτικά εκτεθειμένα άτομα που είναι στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα έλεγα, και εσείς ως βουλευτές είστε στα πλαίσια αυτού του ενισχυμένου κινδύνου. Και υπάρχει και το correspondent banking, δηλαδή πρέπει να ξέρει κανείς τι κάνει με τις ε, τράπεζες τις οποίες είναι κανείς πελάτης και όλες αυτές οι υποχρεώσεις έκαναν τις τράπεζες να συστήσουν συστήματα αρκετά σημαντικά που σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να υπάρχει οργάνωση και υπηρεσία για την πρόληψη του ξεπλήματος βρώμικου με εργαλεία και βάσεις δεδομένων πολύπλοκα για τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, για την ανείχνευση παράνομων δραστηριοτήτων και υπάρχουν και διάφορα εποπτικά και φιλτραρίσματος τέτοιου είδους μηχανισμοί για να δει κανεί εάν έχει να κάνει ενδεχομένως με πελάτη τρομοκράτη αν δεν έχουμε να κάνουμε με παραβίαση κάποιων κανόνων εμπάργου. Πρόκειται λοιπόν για επαχθείς δομές και το ίδιο το σύστημα αυτό είναι αρκετά σημαντικό σε όλες τις τράπεζες. Και βεβαίως υπάρχει η η υποχρέωση να δημιουργούνται βάσεις δεδομένων, να ανταλλάσσονται στοιχεία και ξέρουμε ότι υπάρχει το θέμα την προσωπικών δεδομένων. Πώς να κάνει ανταλλαγή στοιχείων όταν έχει να κάνει με έναν πελάτη ενδεχομένως ύποπτε και συγχρόνως πώς μπορεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη του. Οι τράπεζες δεδομένων είναι ένα άλλο θέμα. Δεν έχουμε κατάλογο των πολιτικά εκτεθειμένων ε, πελατών. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο διαθέτουν οι τράπεζες. Πολλές φορές προσφεύγουν και σε ιδιωτικούς φορείς. Διότι μόνη της μία τράπεζα δεν μπορεί να έχει ε, αρχιοθετημένα όλα τα στοιχεία των πελατών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Επίσης, ξέρουμε πολλές φορές, και αυτό εμφανίζεται στον τύπο, ο, η αναζήτηση αρνητικών στοιχείων για κάποιο πελάτη. Δηλαδή, μήπως ε, έχουν διαρρεύσει στον τύπο κάποια στοιχεία αρνητικά που αφορούν κάποιες δραστηριότητες του πελάτη. Και πρέπει να πω ότι πολλές φορές η αξιοπιστία των στοιχείων που παρέχονται δεν είναι 100% σωστή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω σε εσά τρεις παρατηρήσεις, τρεις επιθυμίες εκ μέρους όλων των ε, τραπεζών της Ευρώπης. Θα θέλαμε σε επίπεδο τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια κεντρική βάση στην οποία να απογράφονται και να καταγράφονται όλες οι εταιρείες με τους δικαιούχους και με τους μετόχους ώστε να έχουμε ένα τέτοιο αρχείο ενιαίο ευρωπαϊκό. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο τις τράπεζες αλλά και τη βιομηχανία και το εμπόριο. Διότι πολύ συχνά δεν έχουμε πληροφορίες και αυτή θα ήταν μια πρώτη επιθυμία εκ μέρους μας, μια ευχή. Αυτό θα μας επέτρεπε και όπως λέγουν και διάφοροι μη κυβερνητικές οργανώσεις, να αυξήσουμε την διαφάνεια. Και πρέπει να πω ότι συμφωνούμε ε, εκ μέρου μα με αυτό το οποίο ζείτε από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τώρα, όσον αφορά για τα άτομα τα οποία είναι πολιτικά εκτεθειμένα, να θέλετε, ξέρω ότι είναι δύσκολο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε έναν κατάλογο ε, συμπεριλαμβάνοντας τέτοια άτομα, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε στις διάφορες χώρες ποια άτομα και σε ποιο επίπεδο ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται άτομα και με ποια χαρακτηριστικά. Στη Γερμανία σε επίπεδο ε, ομοσπονδιακό, σε επίπεδο κρατηδίων. Η προσέγγιση βάση ρισκού θα μπορούσε να γίνει ε, σε επίπεδο κρατών. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει σε επίπεδο Ευρώπης με πιο ομοιόμορφο και ενιαίο τρόπο. Αυτές είναι οι επιθυμίες εκ μέρους ε, της ε, Ομοσπονδίας των Τραπεζών και της Σχετικής Επιτροπής της δικής μου. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε αμέσω τη συζήτηση. Ο εισηγητής, ο κύριος Γιακολίνο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ να αρχίσω από την τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Βόκ. όπου μιλάει για την ευρωπαϊκή προσέγγιση του στον τραπεζικό έλεγχο. Σήμερα μιλάμε για την τραπεζική governance, τραπεζική διαχείριση μέσω της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Οι Γερμανοί όμως θέλουν να βγάλουν από αυτό το δεσμευτικό σχήμα τις συνεταιριστικές τράπεζες. Εσείς πιστεύετε και είναι ερώτησή μου ότι αυτές οι νομοθεσίες μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό φραγμό στο ξέπλυγμα του βρώμικου χρήματος. Τώρα για τον κύριο Στίγκλερ σχετικά με το, σύνδεσμο παρανόμων στοιχημάτων και ανακύκλωσης. Μήπως ε, δεν θεωρείτε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε όλο αυτό το σύστημα είναι η δικαστική και αστυνομική συνεργασία ε, με αμοιβαία εμπιστοσύνη, να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Διότι όταν δεν υπάρχει καμία αντίσταση έναντι αυτού του συστήματος, ε, σίγουρα και βρίσκει ε, και ριζώνει τα παρακλάδια του. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι για να μπορέσουμε εμείς να αντισταθμίσουμε όλα αυτά χρειάζεται συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φαγιόν και παρακαλώ μετά να μας υποδεικνύετε ποιος είναι και ο αποδέκτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω από τον τελευταίο ομιλητή. Είπατε ότι φαντάζεστε ότι σε κάθε χώρα θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό που θα καταγράφονται ή θα δηλώνονται όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αν σας κατάλαβα καλά, αυτό το θεωρείτε και πρώτο βήμα. Το δεύτερο ποιο θα ήταν. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πάμε σε μια κατεύθυνση ότι αυτά τα αρχεία θα διατίθενται και στη δικαστική δικαιοσύνη, στη δικαστική εξουσία, συγγνώμη, θα έχουν πρόσβαση οι δικαστές. Τι να το κάνουμε αυτό το αρχείο αυτή τη στιγμή ε, καταρτιστεί. Ζούμε σε μια περίοδο κρίσης και ε, μιλούμε και για μια φαιά ζώνη που αφορά ε, δικηγόρους, ε, ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές. Και εσείς τι κάνετε εδώ, προτείνετε μέτρα για να εντοπίζονται αυτά τα φύσοπα και να διώκονται και να τιμωρούνται. Κάνετε συστάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Να, έρθω και στα τυχερά παίγνια. Είπατε ότι πρόκειται για ποσά φορολόγητα και προτείνεται να φορολογούνται τα κέρδη. Πώς θα γίνει αυτό και σε πόσα κράτη-μέλη ήδη φορολογούνται ε, τα κέρδη από το Ιντερνετικό στοίχημα. Ο κύριος για την άλλη Ευχαριστώ. Προς τον κύριο Ντελαπιέρ να σας πω ότι χρησιμοποιώ το iPad μου για να βρω ε, περισσότερα στοιχεία για το FIU, τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών και βρήκα ε, στο σελίδα σας FIU.net. Ε, ολόκληρο δίκτυο έχετε στην Ευρώπη και συνεργάζεστε. Πολύ εντυπωσιακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Ωραία, έχετε δίκτυο. Ε, δεν ξέρω, ίσως να μην λειτουργεί τέλεια, γιατί αυτό βλέπω στην ταμπλέτα μου, αυτή την εντύπωση. Εμείς πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για τον κύριο Κώστα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και σας ξανακούω. Είχατε ξανάρθει πριν από λίγα χρόνια και το μήνυμά σας τώρα είναι έτσι ζωφερότερο από ό,τι πριν από ε, λίγα χρόνια που είχατε έρθει. Εμείς πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε γιατί το πρόβλημα είναι σοβαρό, διονγκούμενο και ανισχυτικό. Και για τον καθηγητή Φίτλερ ε, Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ε, να φορολογούνται τα κέρδη από τον Ιντερνετικό ε, τζόγο. Τι γίνεται όμως με τους εθνικούς ε, οργανισμούς λαχείων, κρατικών λαχείων. Εγώ κάθε εβδομάδα αγοράζω λαχείο, αλλά δεν κερδίζω δυστυχώς. τι θα κάνουμε, θα φορολογήσουμε και τα λαχεία. Αν το προτείνουμε αυτό, ε, θα δυσαρεστηθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Οι πολίτες δεν θα αγοράζουν πια λαχεία. Και θα να ρωτήσω και τον κύριο Βακ από τις τράπεζες. Μιλήσατε για άμεσες κυρώσεις και πολύ βαριές. Να πέσει ράβδος. Αλλά ο καθηγητής από το Αμβούργο νομίζω είπε ότι... Υπήρξε μια μεγάλη αμερικανική τράπεζα, δεν ξέρω ποιος το είπε για το Μεξικό και δεν τιμωρήθηκε κανένα υψηλό βαθμό στέλεχος. Και η HSBC κατηγορείται τώρα τι θα κάνουμε, θα τιμωρήσουμε όλα τα στελέχη ή θα βγουν όλοι πεντακάθαροι από εκεί. Τι θα γίνει, δηλαδή θα πάει φυλακή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποργέτσιο για το FT. Να ξεκινήσω με τον καθηγητή Κώστα να τον ευχαριστήσω διότι πολλοί από μας Πολλοί από μας γνωρίζουμε ότι ο καθηγητής παγκοσμίω ε, σε διάφορα θεσμικά όργανα αναφέρθηκε σε αυτούς τους ε, ε, δεσμούς μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και νομίμων ασχολιών. Και εγώ θα συμφωνήσω, θα, θα, θα προσετεριστώ την ερώτηση που ήδη διατυπώθηκε. Και αυτό δηλαδή και λόγω της ε, μεγάλης εμπειρίας που έχει ο καθηγητής στην Αμερική για τη διασύνδεση μεταξύ διακίνησης ναρκωτικών και νόμιμης οικονομίας. Θα ήθελα να μας ε, προσθέσει κάτι για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Διότι Εκεί που φτάσαμε πλέον οι μαθίες φτάνουν στα, ε, στην καρδιά των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να εμποδίσουμε αυτές οι ενέσεις χρηματοδότησης των κρατών προς τις προβληματικές τράπεζες να μην γίνονται ενέσεις προς το έγκλημα. Για τον κύριο Γουάκα, λέει ο μιλητής. Θέλω να ρωτήσω πώς καταφέρνουν οι τράπεζες να μαζεύουν τόσο ακριβείς και αναλυτικές πληροφορίες στο βαθμό δηλαδή που όλες οι τράπεζες, ε, οι περισσότερες τράπεζες που έχουμε στην Ευρώπη έχουν έδρες φορολογικούς ε, παραδείσους όπου ε, κυριαρχεί το, η μυστικότητα και κανείς δεν μπορεί να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα για τον κύριο Φίτλερ θέλω να τον ευχαριστήσω. Ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός γύρω από μια πραγματικότητα, τουλάχιστον για μένα, ε, την οποία ακόμη πρέπει να την καταλάβω. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε ε, και στοιχεία για τα στοιχήματα, για, τα στοιχήματα, αυτό, τα τα, τα, τα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο Και τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε. Διότι διατρέχουμε τον κίνδυνο μαφιόζικης ρήπανσης στον αθλητισμό. Και σε μια χώρα σαν τη δική μου αυτός μέσο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσο, κύριος Γκόμερ, η κυρία Γκόμερ να ερωτήσω τον οποιοδήποτε, αλλά κυρίως τον κύριο Βόκ, το εξή. Στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής κρίσης ακούσαμε ότι οι γερμανικές αρχές έχουν κατάλογο ατόμων με λογαριασμού στο Λίχτενστάιν. Και υπάρχει και στην Ελλάδα ο κατάλογος Λαγκάρντ, η λίστα η στην οποία μπορούν, ε, με την οποία μπορούν οι ελληνικές αρχές να εντοπίσουν ποιους φόρο διαφεύγουν και είναι στους φορολογικούς Πρέπει όμως να πω ότι τα έσοδα από τέτοιου είδους παράνομες και δραστηριότητες είναι σε αμφιβήτηση. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους αρχή. Η... Το Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κεντρική ε, τράπεζα είναι αυτές οι οποίες έχουν εγγυηθεί το κρατικό χρέος των κρατών. Και σημαίνει και στη χώρα μου. Έχουμε την Τρόικα που θέλει να ρυθμίσει το φορολογικό και οικονομικό σύστημα, αλλά πρώτα απ' όλα δεν θέλουν τα άτομα που εντοπίστηκαν στην Ελβετία δεν του ζητούν να επαναπατρίσουν τα κεφαλαία τους και δεν ζητούν και την προέλευση των ε, κονδυλίων που είναι παράμεσα στην Ελβετία. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τα ε, θεσμικά όργανα γιατί δεν κάνουν τίποτα κυρίως για τις χώρες οι οποίες έχουν δοθεί εγγύσεις για την ε, αποπληρωμή του κρατικού στους χώρους. Ευχαριστώ. Κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήμουν μέλος της ειδική Επιτροπής για την χρηματοπιστωτική κρίση εδώ και δώσαμε μαρτυρίες τα άτομα τα οποία έκαναν την έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη στη ΣΥΠΑ, στην Επιτροπή μας και είπε ότι κάποια άτομα και κάποιες τράπεζα όταν επέστησαν την προσοχή στους υπεύθυνου για τα ε, πολύ μεγάλα πτώματα που δόθηκαν και το ότι όλο το σύστημα δεν μπορούσε να φέρει το Ελέγχθη. Γιατί η HCBC. Γιατί. Όταν θα ανακαλυφθεί το όλο σκάνδαλο, ούτε εγώ ούτε εσείς θα είμαστε εδώ. Άρα υπήρχαν άτομα τα οποία ήξεραν τι θα συμβεί. Και πολλά αυτά έχουν σχέση με το γεγονό ότι πιστεύω ότι εδώ, ότι όταν η... Παίρνω το παράδειγμα τη Goldman Sachs. Η Goldman Sachs και η Lehman Brothers αυτά τα χρηματοστικά ιδρύματα όταν είχαν ε, εταιρική, ε, ήταν εταίροι, τους ενδιέφερε η φήμη και μετά δεν τους ενδιέφερε τίποτα. Και τώρα φτάνω στο εξής ερώτημα. Εξετάζουμε τώρα το θέμα των κανονισμών των οικονομικών ελέγχων. Ο Μισελ Μπαρνιέ πρότεινε αρχικά ότι δεν θα πρέπει οι εταίροι στην ίδια εταιρεία να γίνονται ε, για τρία χρόνια οικονομικοί ελεγκτές. Μεγάλη Βρετανία, ο μέσος όρος, ο χρονικός που χρειάστηκε κάποια φορά να γίνει οικονομικός έλεγχος σε μία δημοσιοποίηση ήταν 48 χρόνια. Τώρα προτείνει ο Μισελ Μπαρνιέ 24 χρόνια, μειωθεί ο χρόνος αυτό στο ίμιση. Αρχικά προβλέπαν οι κανόνες ότι θα πρέπει να υπάρχει, ε, όπως είχε αποφασίσει το δικό μας κοινοβούλιο, ε, να υπάρχει η αρχή η οποία να εποπτεύει, όχι να έρχεται μετά για να τιμωρεί. Πιστεύετε εσείς ότι αυτοί που κάνουν τον οικονομικό έλεγχο πέσουν τον δεύτερο ρόλο, δηλαδή δεν κάνουν ε, την εποπτή για να δουν αν όλο κάνουν πάνε σωστά έγκαιρα, αλλά πρέπει εκ των υστέρων να φτάσουν για να δουν ότι κάτι δεν πήγε καλό, όταν ήδη έχει γίνει το κακό. Θα δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές μας. Έχουμε 10 λεπτά. Στις 5 ε, και 20 θα πρέπει να κλείνουμε αυτό το πάνελ. 10 λεπτά λοιπόν. Και παρακαλώ τον δόκτωρα Κώστα μήπως θα μπορούσε να μας δώσει ένα αντίγραφο της τοποθέτησής του. Και σας, παρα... σας το ζητώ προσωπικά ως πρόεδρος αν θα μπορούσατε να μας κάνετε συστάσεις, συγκεκριμένες συστάσεις προς την Επιτροπή μας. Κύριε Ντελεπιέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση αφορά στο EFIU NET. Η Financial European Unity έχει ένα δίκτυο, ένα πληροφορικό δίκτυο το οποίο έχει ε, στηθεί, λειτουργεί και μας επιτρέπει να διαπιστώνουμε εάν γνωστοί οργανισμοί στο Βέλιο βρίσκονται σε μια άλλη χώρα της ένεσης. Πρόκειται για ένα σύστημα data matching. Άλλες δυνατότητες επίσης μελετάμε σήμερα. Υπάρχει μια πλατφόρμα και στην ε, Κομισιόν που παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται το IFAUNet. Ε, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία θέλησαν μέσω του IFAU να κρατήσουν μια λογική σειρά. Έχουμε στα δικαστικά την Eurojust, την Europol για τα αστυνομικά θέματα Υπάρχει ένα σύστημα οδηγιών ε, για την πρόληψη της λεύκανσης με κεντρικό σημείο της FIU και η αρχική ιδέα ήταν να πούμε να μην έχουμε επικάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα μέσω του FIUNET η λύση της Επιτροπής, είναι, της Κομισιόν δηλαδή, είναι να ενταχθεί το net μέσα στην Europol και αυτό για να την αξιοποίηση, τη λογική αξιοποίηση των μέσων. Ε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές ΑΙΦΑΙΟΥ έχουν δεχτεί την πρόταση, αλλά παραμένουν πεπισμένες ότι Ιδανικό θα ήταν, ε, επειδή έχουμε πολλές οδηγίες για ε, την ε, λεύκανση του ευρωπαϊκού χρήματος, ότι θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν πέρα από τα εθνικά FIU μία ευρωπαϊκή δομή υψηλού επίπεδου, όχι μόνο για να προχωρήσουμε σε λειτουργικό επίπεδο, αλλά και για να προχωρήσουμε στη στρατηγική ανάλυση του κινδύνου λεύκανσης και να απαντήσουμε και σε μία από αυτές τις νέες συστάσεις. Δηλαδή να έχουμε μία αιτήσια αξιοποίηση του κινδύνου των απειλών όπως εκφράζονται σε κάθε κράτος μέλος. Και Σχετικά τώρα με τους ελεγκτές, Οι πληροφορίες που μας έρχονται από τις τράπεζες είναι πληροφορίες που δεν προχωρούν ποτέ μακρύτερα από αυτό που οι ελεγκτές μπορούν να έχουν κατά τη διάρκεια της αποστολής τους. Γι' αυτό λοιπόν οι ελεγκτές συμπεριλαμβάνονται μέσα στο ίδιο το σύστημα των δηλώσεων και πρέπει να κάνουν δηλώσεις ε, ε σχετικά στην FAU. Υπάρχει έλεγα αυτή η υποχρέωση, αλλά διαπιστώνουμε ότι μέγα μέρος αυτών των ελεγκτών δεν κάνουν δηλώσεις στα πλαίσια της εφαγιού. Και αυτό σας το λέω γιατί είναι, ένα όντως, είναι όντως ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αναλύσουμε, δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση αυτών των ανθρώπων στην όλη διαδικασία ελεύκανσης του βρώμικου χρήματος. Κύριος Κώστα. Πάρα πολύ σύντομα ε, να απαντήσω και στην ερώτηση ε, της Προέδρου του κυρίου Νιουτοντάν και του κυρίου Μποργέζιο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα Έχουμε δει στοιχεία. Εκατέρωθαν το Ατλαντικού σε πολύ μεγάλες χώρες. Ότι οι αρχές, οι ρυθμιστικές, οι κυβερνήσεις και τα δικαστήρια και οι τρεις στην επιβολή κυρώσεων δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το πρόβλημα του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Σας μίλησα για 430 εκατομμύρια ε, δολάρια στην Αμερική χωρίς πρόστιμο, χωρίς καμία επίπτωση. και έγινε όταν ήταν στο η οικονομική κρίση μετά τους Lehman Brothers. Το αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα δεν μπορούσε να αντέξει την κατάρρευση μιας άλλης μεγάλης τράπεζας. Και το α, συγκάλυψαν, ας πούμε. Η ιστορία θα δείξει τι έγινε και τι έπρεπε να γίνει αν θα έπρεπε να τιμωρηθούν οι άνθρωποι. Ένα μεταξύ δύο κακών το μη χείρον βέλτιστον. Περισσότερες ρυθμίσεις και κανονισμοί προτάθηκε αυτό και από το προηγούμενο πάνελ. Ακούσαμε Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία συναλλαγή όταν είναι άγνωστος προς την τράπεζα ο κομιστής ή ο πελάτης. Είδαμε πόσο εύκολο είναι και πόσο επιπόλαιο ε, να γίνει. Ε, δεν λειτουργούν τέτοιες ρυθμίσεις σαν αυτές που υπάρχουν. Εντάξει, θέλετε περισσότερες ρυθμίσεις, αλλά δεν ξέρω αν αυτές θα αποφέρουν αποτελέσματα. Τι θα πρέπει όμως να κάνουμε γι' αυτό αυτό που χρειάζεται και αυτό είναι ο δικός σας ρόλος των Ευρωπαίων νομοθετών θα πρέπει να αναγκάσουμε τις τράπεζες να επιστρέψουν στην καταγωγή τους. 500 χρόνια οι τράπεζες ήταν το βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας. Τώρα το έχουν γυρίσει και έχουν γίνει καζίνα. Έχουν γίνει τόπος τζόγου οι τράπεζες. Για τους καταθέτες ε, και καταθέτουν τα χρήματά τους και τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για το λάθος τρόπο. Εάν ε, και σκοπό. Εάν δεν αναγκάσουμε τις τράπεζες να αλλάξουν τακτική, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το πράγμα και εσείς οι νομοθέτες να κάνετε ε, νόμους και το κοινό, το ευρύ κοινό, οι πελάτες ας πούμε, θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ότι όποια τράπεζα δεν συμμορφούνται και παραβιάζει τα βασικά στοιχεία θα πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες του νόμου. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Δύο λεπτά ο κύριος Φίτλερ και άλλα δύο μετά ο κύριος Βακ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ε, επιβολή του νόμου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία συνεργασία. Και ο τζόγος και το οργανωμένο είναι θέμα για το οποίο σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει και διεθνώς να υπάρχει συνεργασία. Και πολλά θα κερδίσουμε αν συνεργαστούμε όχι μόνο σε περιφερειακό και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο αλλά και μεγαλυστή των διαφόρων τμήματων των διαφόρων οργανισμών. Πιστεύω ότι υπάρχουν προφορίες που θα ήταν χρήσιμες για τους άλλους χρήσιμες προφορίες που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό λοιπόν είναι τελικά κάτι στο οποίο θα πρέπει να προσβλέψουμε όσον αφορά τους φόρους και τον τζόγο. Θα αρχίσουμε τη δική σας ερώτηση. Ξέρουμε ότι όλα αυτά ε, τα θέματα της λοταρίας είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δαπανερό και κανένας δεν θα τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Τώρα όσον αφορά τα, ε, το τζόγο τον ηλεκτρονικό, επίση είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Για να κάνει κανείς ε, ε, ξέπλυμα, να μπορέσει να καταπληρώσει το ξέπλυμα χρήματο δεν χρειάζεται να φορολογήσει. Τώρα, τα λαχεία. Αν υπάρχει μία χώρα που δεν φορολογεί ε, τον ε, τζόγο, όλοι εκεί θα πάνε. Αν το κάνει αυτό η Γερμανία, εκεί θα πάνε όλοι. Και αν οι άλλοι το... Δεν ξέρω τώρα ποιος θα φορολογεί, δεν ξέρω ποια χώρα το κάνει αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος είναι αυτός που δεν φορολογεί. Γερμανία. Όσον αφορά τα ε, στοιχήματα και το ξέπλυμα χρήματος. Αυτό αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δραστηριότητα. Τα στημένα παιχνίδια είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει μόνο στο ποδόσφαιρο στην Ιταλία, αλλά παντού στην Ευρώπη. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η αγκαιριότητα τον δεν είναι κάτι το οποίο λάμπει. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Επίσης, με το τζόγο online, τον ηλεκτρονικό πολλά γίνονται. Διότι έχουμε να κάνουμε μια τεράστια αγορά. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ξεπερνιούνται τα όρια. Τέλος πάντων, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Η πρώτη αφορά τι θα ανάξει η Τραπεζική Ένωση και η διαχείριση σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας με ρυθμιστική αρχή σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του έχω, αυτό θα αφορά κυρίως τους ε, οικονομικούς ε, ε, κινδύνους και τα, τους ιδίους πόρους. Όσον αφορά την ρύθμιση σε θέματα πρόληψης του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, αυτό θα αφορά κυρίως τις χώρες, ακόμη και με την Τραπεζική Ένωση. Δεύτερη ερώτηση Μιλήσατε για τι ε, τράπεζε δεδομένε και τι πληροφορίε που διαθέτουν οι τράπεζε. Έχουν πάρα πολλέ πληροφορίε οι τράπεζε, δεδομένου ότι όλε οι τράπεζε ελέγχουν όλες τις ε, διεθνεί του συναλλαγές για να μην χρηματοδοτείται η τρομοκρατία και να επιβάλλονται κλειώσει. Όλες τις δραστηριότητες των πελατών του ελέγχουν θέσατε το ερώτημα το μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή τέτοιου πληροφοριών. Δυστυχώ, έτσι όπω έχουν τα πράγματα και σύμφωνα με του κανόνε, δεν μπορεί μια τράπεζα να ανταλλάξει τέτοιου πληροφορίε παρά μόνο με μια άλλη τράπεζα όταν πρόκειται για συναλλαγή που αφορά τι δύο τράπεζε. Και απαγορεύεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων με ε, λογιστέ, με δικηγόρου κτλ. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω. Στη χώρα μου, στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με την ρυθμιστική αρχή για τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, τον τζόγο των ηλεκτρονικών. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι να μπορέσουν να ανοιχνεύσουν τα παράνομα sites, όπου έχουμε πάρα πολλά sites τα οποία είναι νόμιμα, αλλά πάρα πολλά τα οποία είναι παράνομα. Εκεί διακινείται μεγάλο χρήμα και κανείς δεν μπορεί να τα ανοιχνεύσει εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε το μέσο που θα μας επιτρέψει να ανοιχνεύσουμε αυτά τα παράνομα sites και όταν θα τα διαλύσουμε πώς θα αποφύγουμε να μην ξαναεμφανιστούν με άλλη ονομασία. Είναι ένα σχέδιο το οποίο, με το οποίο ασχολούμαι εγώ προσωπικά. Τώρα, πώς έχουν πληροφορίες για τις διάφορες εταιρείες που εδρεύουν στους ε, φορολογικούς παραδείσους η τράπεζες. Εάν δεν δώσουν κάποιες πληροφορίες δεν μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους. Εάν μια εταιρεία ή κάποιος έρχεται εκ μέρους μιας εταιρείας η οποία είναι καταγεγραμμένη σε ένα φορολογικό παράδεισο να ανοίξει λογαριασμό σε μια τράπεζα, το καταστατικό της τράπεζας δεν έρθει. Πρέπει να ξέρει βάσει πιστοποιητικού ποιος είναι ο αποδέκτης, ο δικαιούχος. Και λέει και τον κάφιο ότι δεν μπορεί κανείς ως τράπεζα να έρθει σε επαφή αν δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Τώρα, τελευταίο ερώτημα, τα φορολογικά προβλήματα, φοροδιαφυγή και οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο Λίχτενστάιν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη σε παγκόσμιο, πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί της ε, φοροαπάτης. Συνοπτικά έχετε το πρώτο επίπεδο απόκρυψη φορολογικών στοιχείων. Κάποιος ο οποίος ερχάζεται και αποκρύπτει από την εφορία ένα μέρος των δραστηριοτήτων του που του αποφέρουν. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Μετά έχετε την ε, φοροδιαφυγή. Δηλαδή όχι μόνο αποκρύπτετε τα έσοδα που έχετε, αλλά τα πάτε στην Ελβετία τα κέρδη Τώρα, το cash pooling, αντί να το έχει μια εταιρεία στην Πορτογαλία, είναι πορτογαλική, το πάει στην Ελβετία. Και εάν το cash management, η διαχείριση λοιπόν του ρευστού μιας επιχείρησης είναι στην Ελβετία, δύσκολα μπορεί κανείς να ξέρει τι γίνεται. Και στο τέλος υπάρχει και η φοροαπάτη, δηλαδή ζητάει κανείς βάσει λανθασμένων και πλαστών εγγράφων να του αποδοθεί το ΦΠΑ από το κράτος, το οποίο δεν έχει καταβάλει. Πρόκειται λοιπόν για οργανωμένη ε, απάτη και ξέρουμε ότι στην Ιταλία ε, υπήρξαν κάποιο τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις φοροαπάτης. Είναι το τρίτο επίπεδο. Δεν ξέρω αν απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά ξεπέρασε τα δύο λεπτά που μου είχαν δοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την για την ποιότητα των επιχειρημάτων. Τώρα παρακαλώ πριν ολοκληρώσουμε να έρθει εδώ ο κύριος Κροτσέτα στο Προεδρείο, διότι όπως ε, σας ε, προανήγγυλα, ο συνάδελφος το προηγούμενο Σάββατο έγινε πρόεδρος της ε, Σικελίας, της περιφέρειας Σικελίας. Θα είναι η τελευταία τοποθέτηση του Ροζάριου ως Αντιπροέδρου και μέλους ε, της Επιτροπής μας. Παρακαλώ Ροζάριο. Allora, Rosario, io πριν σου δώσω το λόγο, Θα ήθελα να σου πω το εξή. Ήμασταν στην Ιταλία εμείς. Πήγαμε στο Μιλάνο, στο Παλέρμο και στην ε, Ρώμη. Οι συνάδελφοι εξεπλάγησαν μερικά πράγματα θετικά αλλά για άλλα αρνητικά σχετικά με αυτά τα οποία είδανε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες συστάσεις για τις οποίες θα συμφωνήσουμε. Συναντήσαμε την Μιχτή Επιτροπή ε, κατά της μαφίας ε, στην Ιταλία και συνεδριάσαμε από κοινού. Εγώ την Παρασκευή πήγα στην εισαγγελία του Τράπανη και συνάντησα το Δημοτικό Συμβούλιο, είδα τους ε, εισαγγελείς, ε, τους δικαστές και τα μηνύματα που στάλθηκαν είναι πολύ αρνητικά. Λοιπόν, εγώ απευθύνω αυτές τις εκκλήσεις προς εμάς, ε, διότι έχουμε την κοινή ιστορία. Ξέρω την ευαισθησία σου προς γι' αυτά και σε παρακαλώ να επαγρυπνείς. Και η Επιτροπή μας προφανώς συμφωνεί. Σε παρακαλώ με παγρυπνείς για τη χρήση των κονδυλίων της, της χρηματοδότησης Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα παραγράφησαν αδικήματα τα οποία παρέγραψαν στην Σικελία, στη, χώ, στη γη μας δηλαδή, 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια ευρώ κοινωνικά κονδύλια παραγράφησαν. Για το θέμα των, ε, δημο, των ε, δημοπρατήσεων. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι συνάδελφοι με άκουσαν και ακούσαμε διάφορους μάρτυρες στα δικαστήρια και ξεπλάγησαν εξεπλάγησαν από τις προσωπικές ιστορίες. Ε, ε, έχουμε πολλούς ε, τέτοιους μάρτυρες στην, στη Σικελία. Χθες ένας έκανε μια πολύ ισχυρή δήλωση, ο Μαρσέλου Κουτρό. Ακούσαμε επίσης και τα μέλη των οικογενειών θυμάτων της Μαθίας. Εγώ άκουσα διάφορους άκουσα άτομα τα οποία, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των αγαθών της, ε, που έχουν κατασχεθεί από τη μαφία. Και μου ανέφεραν ότι με δυσκολία μπορεί κανεί να διαχειριστεί την ε, μαφιόζικη περιουσία, με δυσκολία γίνεται ανταγωνιστική διαχείριση τη διαχείριση. Και ζητούν από εμά να ρυθμίσουμε όλα όσα δεν λειτουργούν μέχρι σήμερα. Τελευταία έκκληση που σου απευθύνω και που σίγουρα και εσύ συμμερίζεσαι είναι η έκφραση της υποστήριξής μας και της υποστήριξής σου προς τις εισαγγελίες και τους εισαγγελείς που είναι στην πρώτη γραμμή. Εμείς ακούσαμε ένα σωρό κατά τη διάρκεια της ακρόασης και είμαι πεπισμένος ότι η δική σου υποστήριξη δεν θα τους λείψει. Σου δίνω λοιπόν το λόγο ολοκληρώνοντα και η Επιτροπή μας σίγουρα θα και εξετάζει προσεκτικά του σύνεγγυ τη δουλειά της Επιτροπής Αντιμάφια στην Σικελία. Διότι έχουμε απόλυτη σύγκληση προθέσεων κύριε Κροτσέτα. Καλησπέρα σε όλους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση τοποθετούμε σε αυτήν την ε, επιτροπή, διότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα παραιτηθώ για να ασκήσω το λειτουργήμά μου ως πρόεδρος της Σικελίας. Η Σικελία από τον, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά είναι για πρώτη φορά ε, που εκλέγει κάποιον ο οποίος είναι σαφώς τοποθετημένος κατά της μαφίας. Πρόκειται για κάτι το ιστορικό μέσα στα κοινωνικο-πολιτικά δρόμενα της περιοχής, της περιφέρειας. Και μιλάω εδώ για την άμεση εκλογή από τους πολίτες. Μία περιφέρεια όπου 8 πρόεδροι της περιφέρειας από τον μεταπόλεμο και μετά πήγαν φυλακή. Και οι δυο ε, απομακρύνθηκαν λόγω σχέσεων με τη μαφία. Η εκλογή μου λοιπόν δεν ήταν καθόλου απλό πράγμα και καθόλου απλό πράγμα και η δουλειά που με περιμένει δεν είναι ιδιαίτερα ισχύ. Πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, θα πέσει φαρμάκι, γουρσουζιά, ε, τέλο πω μεγάλες δυσκολίες και εγώ θα προσπαθήσω να ε, υπερασπιστώ την αξιοπρέπεια του σικελικού λαού. Θα παρακολουθούμε από κοντά το τι διαμείβεται στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα σε αυτή την Επιτροπή, ούτω ώστε να έχουμε ισχυρά κείμενα τα οποία θα έχουν τη συνέστηση ότι η μαφία δεν είναι απλά ένα πρόβλημα της Σικελίας ή της Ιταλίας, αλλά ε, έχουν παγκοσμιοποιηθεί οι μαφίες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Ιούλιο του 2004 με ένα ένταλμα συλλήψεων στην Τζέλα αρχαία γέλα όπου το ένταλμα αφορούσε έναν σικελό μαφιόζο και έναν λιθουανό μαφιόζο, ο οποίος είχε μάλιστα αναλάβει την εντολή να με καθαρίσει. Βλέπετε λοιπόν η μαφία σήμερα απευθύνεται σε αλλοδαπούς κίλερ. Δείτε πώς αλλάζει ο κόσμος, πώς εξελίσσεται αλλά το, ε, το πιο εντυπωσιακό ήταν στις 6 Δεκεμβρίου του 2003. Αυτό το τηλεφώνημα το οποίο ε, έπιασε η αστυνομία εκτός από το να παζαρεύουν τη ζωή μου αυτό το οποίο μου δημιούργησε ρίγη ήταν το εξής που έλεγε στις 12 Δεκεμβρίου του 2003 θα έχουμε μία συνεδρίαση στις Βρυξέλλες και από τις αποφάσεις αυτής της Επιτροπής εξαρτώνται μεγάλες αποφάσεις για τη Σικελία και τη Λιθουανία. Δηλαδή πολλά σήμαινε αυτό για τη Σικελία και για τη Λιθουανία, για τις μαφίες τους και πήγα να δω τι γινόταν τότε και ήταν η συνεδρίαση της ε, διάσκεψης κορυφής όπου αποφάσισαν την είσοδο της Λιθουανίας στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν εμείς να σκεφτούμε πώς οι μαθίες εδώ και καιρό έχουν επιτεθεί κατά των και έχουν παγκοσμιοποιηθεί, ενώ η πολιτική ακόμη με δυσκολία σήμερα μπορεί, ε, καταλαβαίνει όλη αυτή την αλληλοδιασύνθεση των μαφιών. διεθνώς και τις διαθέσεις που έχουν οι μαθίες με τα θεσμικά όργανα. Όταν εμείς μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ε, φως φανάρι, δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μαθία της Σικελίας. Διάφορες ε, χώρες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η τοπική μαφία διαχειρίστηκε τα κονδύλια. Αυτό Είπαμε λοιπόν η Σικελία, η μαφία δεν είναι περιορισμένη μόνο σε μία χώρα. Διότι όσο η μαφία ήταν ε, απλά και μόνο εγκληματικό φαινόμενο ή στρατιωτικό φαινόμενο έφτανε. Μπορούσε κανείς να τη χτυπήσει στην επικράτειά της. Αλλά σήμερα η μαφία λειτουργεί και χωρίς τον έλεγχο της επικράτειας. Για να προχωρήσει κανείς το έγκλημα στο παρελθόν χρειαζόταν ένα στρατός για να εγκληματίσει. Ένας Ιταλός μελετητής έχει θεωρητικοποιήσει την, την ύπαρξη μιας μαφίας χωρίς μαφιόζους. Μπορούμε να έχουμε μαφιόζικα φαινόμενα χωρίς να υπάρχει το εγκληματικό ή στρατιωτικό σκέλος στη μέση διότι τα επίπεδα διαστροφής ε, τα οποία έχουν, ε, στα οποία έχει φτάσει ο κόσμος της οικονομίας, ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ανοχή, η άγνοια όλων αυτών των διαδικασιών από, τα θεσμικά, από τους θεσμούς δημιουργεί έναν underground κόσμο, έναν υπόγειο κόσμο όπου κινείται η οικονομία γενικά και κάποια μέρα ανακαλύπτεις εσύ ότι ψάχνεις τη μαφία ε, στη Σικελία και τελικά κοίτα να δεις εδώ στην, σε μια πλατεία στις Βρυξέλλες έκαψαν ένα εστιατόριο, πυρπόλησαν ένα εστιατόριο και οι τεχνικοί μετά θα πούνε ότι επρόκειτο για αυτό πυρπόληση, το ίδιο πράγμα που γίνεται και στο Παλέρμο. Όπου βέβαια στο Παλέρμο πολλές φορές αυτή η πυρπόληση είναι θέμα το ότι δεν πληρώθηκε, δεν, πληρώθηκε η δόση του εκβιασμού, αλλά αναρωτιέμαι τι γίνεται με τα... Πού πάνε τα λεφτά της διακίνησης όπλων, ναρκωτικών κλπ. 170 δις ευρώ το χρόνο είναι τα κέρδη της μαφίας στην Ιταλία και 400 δις στην Ευρώπη. Μα πού πάνε αυτά τα λεφτά, δεν πάνε κάτω από τα στρώματα. Έχουμε και τα 70 δις από τη διαφθορά στην Ιταλία και 200 κάτι στην Ευρώπη. Πού στο καλό πάνε όλα αυτά τα λεφτά Το τραπεζικό σύστημα έχει και αυτό το ρόλο του στην παράνομη διαχείριση. Τώρα, στη, μένα προσωπικά σας λέω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια που θα είμαι πρόεδρος θα χτυπήσουμε τη μαφία άνευ προηγουμένου. Η Σικελία δεν θα θεωρείται πλέον η περιοχή της μαφίας, αλλά η πιο προωθημένη περιοχή για την καταπολέμηση της μαφίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέτρα για τη διαχείριση των δημοπρασιών, τον έλεγχο των επιχειρήσεων, λίστα των επιχειρήσεων, is white list ε, των επιχειρήσεων που μπορούν να συνεργαστούν με το, με το δημόσιο, ε, σοβαρούς ελέγχους ε, κατά της μαφίας. Αλλά αυτά τα μέτρα δεν θα έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα αν τελικά ας πούμε η και επιχείρηση που δεν μπορεί να εργαστεί στο Παλέρμο ή στην Κατάνια θα πάει στο Βερολίνο ή στο Παρίσι διότι εκεί δεν υπάρχουν τέτοιου, τέ, τέτοιοι έλεγχοι. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπόψη μας ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο είτε θα ε, αγωνιστούμε αποτελεσματικά και ότι αυτό μας αφορά όλους ή αλλιώς δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Εγώ θα ήμουν έτοιμος να έχουμε και μία σύμβαση, μία σύμβαση με την ε, Επιτροπή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα database ε, των ε, δημοπρατήσεων ε, μια, ένα παρατηρητήριο για την, ε, στην Σικελία για την αστυνομία και την εισαγγελία και να είμαστε η πρώτη χώρα η οποία κάνει κάτι τέτοιο. Θα κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν μπορούμε να αγωνιστούμε κατά της μαφίας σε μία και μόνη χώρα. Και αυτό όχι γιατί οι μαφιόζοι έχουν πάει παντού, αλλά γιατί σε όλες τις χώρες δεν έχουμε μόνο τις μαφίες που έρχονται από άλλες χώρες. Υπάρχουν και οι aborigines μαφίες, οι ενδογενείς μαφίες, οι οποίες λειτουργούν με το ίδιο σύστημα της Κόζα Νόστρα. Πρέπει λοιπόν εμείς να διαλύσουμε την Κόζα Νόστρα. Έχουμε παγκοσμιοποίηση του συστήματος Κόζα Νόστρα. Το μοντέλο Κόζα Νόστρα είναι το εγκληματικό μοντέλο του, της τρίτης χιλιετίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πρέπει να ξεκινήσουμε μια νέα μάχη, έξυπνη μάχη και ελπίζω αυτή η Επιτροπή την οποία θελήσαμε ιδιαίτερα να μπορέσει να μας δώσει ένα αληθινό και ειλικρινές αποτέλεσμα αφήνοντα κατά μέρος της προκαταλήψεις για την προάσπιση πολιτικών ή εθνικών συμφερόντων. Εδώ δεν είναι θέμα η πολιτική, μια πολιτική επιλογή ή μια άλλη. Το θέμα είναι αν θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικό μέλλον ελευθερίας στην Ευρώπη και αν θέλουμε η παλιά ε, δημοκρατική και φιλελεύθερη Ευρώπη να έχει ένα μέλλον ή αλλιώς ε, τα υπόγεια εγκληματικά λόμπις ε, να διαχειρίζονται την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Πολλές ευχές. για την εντολή σου. Παρακαλώ τώρα να φύγετε για να ξεκινήσουμε με ένα τέταρτο καθυστέρηση τη συνεδρίαση των συντονιστών. Η επόμενη συνεδρίαση 28 Νοεμβρίου από τις 9 στις 12 και μετά από τις 15 μέχρι τις 18 και 30.